ότι την τελευταία φορά που είχαμε ε, τον Chief Negotiator, τον σε διαπραγματευτή, ήταν τον Ιούλιο, αν, αν, δεν κάνω λάθος. Χαίρομαι πάντως που σας ε, ξαναέχουμε. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε ε, λίγο πρόβλημα και χρειάστηκε χρόνος έτσι ώστε να εγκριθούν οι ε, εντολές και ε, ε, αμέσως μετά τέλη Μαΐου, οπότε και είχαμε τις εντολές, ε, ξεκινήσαμε τις διαδικασίες με τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία. Μάλιστα ξεκινήσαμε στην Καμπέρα με, για το ξεκίνημα των διαπραγματεύσεων με, τους, με την Πρωθυπουργό και τον τότε Υπουργό Εμπορίου. Ήταν μια, και με τον Επίτροπο φυσικά, ήταν μια πάρα πολύ καλή έναρξη διαπραγματεύσεων και από πλευρά της Κομισιόν και ε, η αίσθηση γενικά για τον πρώτο γύρο ήταν πάρα πολύ ε, καλή. Αυτός ο γύρος έγινε ε, στις Βρυξέλλες από τις 2 μέχρι τις 6 Ιουλίου. Στον πρώτο γύρο είχαμε 17 ομάδες εργασίας. Πολλές από αυτές αφορούσαν ανταλλαγή απόψεων και επεξήγηση των ε, στρατηγικών ε, της κάθε ε, πλευράς. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα εκτός από τις διατάξεις, τις γενικές θεσμικές διατάξεις. Επίσης, προσπαθήσαμε έτσι ώστε να έχουμε έτοιμες και στο τραπέζι ε, της ε, προτάσεις ε, γιατί είχαμε αργήσει όσον αφορά το θέμα των εντολών άρα θέλαμε να μπούμε στην ουσία αμέσως. Η αυστραλιανή πλευρά έχει υποβάλει τρία κείμενα εμείς είχαμε δώδεκα. η αυστραλιανή πλευρά τρία έγιναν συζητήσεις όμως ε, τα κείμενα της Αυστραλίας ήρθαν αρκετά ε, αργά, αλλά δεν μπορούσαμε να έχουμε πολλές επεξηγήσεις. Σε πάση περιπτώσει, ξέρετε ότι έστω και με αυτούς τους όρους οι συζητήσεις είναι πάντα πάρα πολύ χρήσιμες, γιατί οι εμπειρογνώμονες ε, καταφέρνουν να δουν πού βρισκόμαστε, έστω και αν δεν μπορούμε πλήρως να ασκήσουμε, την, να προχωρήσουμε τη συζήτηση. Έγινε λοιπόν οι πρώτες βασικές συζητήσεις ε, για ε, αυτήν την διαπραγμάτευση. Σε γενικές γραμμές πρέπει να πω ότι η συζήτηση έγινε σε πνεύμα ανοιχτό και με καλή έτσι, χημεία μεταξύ των ε, διαπραγματευτών. είναι επαγγελματίε διαπραγματευτέ από πλευρά και τη Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και επομένω θα προχωρήσουμε καλά ταυτόχρονα και έστω και αν υπάρχει αρκετή σύγκληση σε πολλά κεφάλαια. Ξέρουμε από το πρώτο σκόπινγκ ότι βεβαίως υπάρχουν και κάποιες, ε, ε, κάποια πεδία πιο προβληματικά. Τα γνωρίζουμε τώρα. Βεβαίως έχουμε θέματα πολύ ευαίσθητα όσον αφορά την, ε, την γεωργία ζάχαρη και βόιο, επίσης τις ε, γεωγραφικές ενδείξεις και αυτές μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα. Ήδη έχουμε για το φθινόπωρο ένα πολύ φιλόδοξο ε, πρόγραμμα με ε, βίντεο διασκέψεις, τηλεδιασκέψεις. Και περί τα ε, του Σεπτέμβρη, τη βδομάδα της 24 η ε, θα έχουμε τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Αυστραλίας ε, εδώ για συνάντηση και μαζί μου, όπου θα λάβουμε υπόψη μας την έκβαση όλων των τηλεδιασκέψεων. Μετά θα ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων την εβδομάδα της 19ης Νοεμβρίου. Και αυτό θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Σε γενικές γραμμές ε, τα πράγματα ξεκίνησαν καλά, ως, άλλοτε, ως άλλωστε ανεμένετο. Ε, είχαμε καλές συναντήσεις στην ε, Καμπέρα, είχαμε μια καλή συνάντηση και με τους επικεφαλείς διαπραγματευτές το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Ίντα ε, μας ε, υποστήριξαν και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Πρόκειται για μια σημαντική διαπραγμάτευση γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν εταίροι ε, που έχουν μερική πρόσβαση. Έχουμε επίσης πολλά πεδία επί των οποίων μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο έτσι ώστε να αναπτύξουμε τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου, τις FTAs και οπωσδήποτε, λαμβάνοντα υπόψη τις παρούσες συνθήκες στο διεθνές εμπόριο, θα δώσουμε με αυτόν τον τρόπο αυτό ένα, ε, ένα μήνυμα ότι πιστεύουμε στις ε, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, ε, ότι προχωρούμε και αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκε, είναι κάτι εξαιρετικά θετικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Μόσορ, τον εισηγητή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τη βασική διαπραγματεύτρια. Είναι πολύ καλή η ώρα για αυτή τη συζήτηση μετά τον πρώτο γύρο και επειδή τώρα το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο θα γίνει το, η εργασία μεταξύ των συνόδων. Όπως είπε η κυρία Διαπραγματεύτρια, είναι αλήθεια ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισήμως ε, και επανειλημμένα τρεις φορές σε τρία επίσημα ψηφίσματα, διαφόρων ειδών ψηφίσματα, έδειξε ισχυρή υποστήριξη των διαπραγματεύσεων με έναν πολύ σημαντικό για μας εταίρο. Ε, υπάρχουν κάποια ε, περιορισμοί, κάποιοι όροι, ε, αλλά αυτό δεν περιορίζει την Αυστραλία. Αυτό είναι μεγάλη ευκαιρία για μας να ξεπεράσουμε κάποιες παραδοσιακές αντιλήψεις, ε, μονόπλευρες αντιλήψεις για τη γεωργία που είχαμε παλιά σε εμπορικές σχέσεις, αν και βέβαια η γεωργία παραμένει πολύ σημαντικό θέμα στις διαπραγματεύσεις. Επίσης ε, αξίζει να σημειώσουμε και αυτό το είδα και στο παρελθόν μου, με τις μεταρρυθμίσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σύγχρονος παίκτη στη Γεωργία που έχει ξεπεράσει τα παλιά κλισέ. Χαίρομαι που μπορώ να τονίσω ότι υπάρχει μεγάλη ισχυρή στήριξη των διαπραγματεύσεων από την επιχειρηματική κοινότητα και εδώ και, και στην Αυστραλία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε μια αντιπροσωπεία ε, με επικεφαλή στον Σερ Πίτερ Κόστρο που ε, ε, εξεδήλωσε την υποστήριξη στις διαπραγματεύσεις και αυτό ισχύει και για την ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα που συναντούμε συχνά. Φιστώ την προσοχή σε όλους στις διαπραγματεύσεις, στις διαβουλεύσεις με τη βιομηχανία που συνεχίζεται μέχρι 7 Σεπτεμβρίου και οργανώθηκε από την Κομισιόν. Ευχαριστούμε. Ε, ενθαρρύνω τη βιομηχανία να συμμετέχει γιατί αυτό θα βοηθήσει και την Κομισιόν και ε, την άλλη πλευρά στις διαπραγματεύσεις. Ένα ερώτημα είναι πότε θα, έρθουν τα, θα δημοσιευτούν τα αποτελέσματα από την συνεχιζόμενη ανάλυση. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Ε, δηλαδή πρέπει να έχουμε πρόσβαση στις αναλύσεις και ε, αξιολογήσεις που έγιναν από την Κομισιόν το ταχύτερο δυνατό. Θα γνωρίζετε ότι η έκθεση του πρώτου γύρου δείχνει ότι υπάρχει αποφασιστικότητα και επαγγελματισμό. Ε, η διαρευνητική διαδικασία ήταν πολύ καλή, γνωρίζονται οι δύο πλευρές, ξέρουν προτεραιότητες, ευαισθησίες, οπότε όλα αυτά είναι καλά υλικά για μια στέρεη πρόοδο και ταχεία πρόοδο. Υπάρχουν και δύσκολοι τομεί. Προφανώ ε, γι' αυτό γίνονται διαπραγματεύσεις η πρόσβαση για την Αυστραλία στην ε, γεωργική αγορά, ε, γεωγραφικές ενδείξεις, ε, δημόσιες συμβάσεις και σε κεντρικό επίπεδο, κανόνες SPS και ενία στήριξης και ένα θέμα αν οι λύσεις αρχίζουν να διαφαίνονται σε κάποιο βαθμό. Καλό είναι να προχωρήσουμε γρήγορα για να έχει νόημα, όπως είπε το περασμένο φθινόπωρο Γιούγκερ. Ε, έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα. Στις 19 Νοεμβρίου είναι ο δεύτερο γύρος. Οι επίσημοι γύροι έχουν μεγάλο μεσοδιάστημα, αλλά ε, μπορούμε να το δούμε και πριν από το τέλος της Κομισιόν καλό θα ήταν να ε, υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Πότε θα περιμένουμε ανταλλαγές, οι πρώτες ανταλλαγές προσφορών, πότε θα γίνουν οι ανταλλαγές. Ε, η παράλληλη διαδικασία της εμπορικής πολιτικής και του σχετικού διαλόγου που κατάλαβα ότι γίνεται back to back αν θέλετε και έχει και μια διμερή διάσταση εκτός από την πολυμερή και ε, ε, δεν ξέρω ακριβώς Πώς θα συνεχιστούν δύο διαδικασίες, θα παραμείνουν χωριστές, θα επικαλύπτονται σε ένα βαθμό οι δύο διαδικασίες. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν το έχω ξαναδεί σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις αυτό. Τέλος σημαντικό όμως, οι πρόσφατες πολιτικές αλλαγές ε, στην Αυστραλία και αν θα επηρεάσουν τα χρονοδιαγράμματα των διαπραγματεύσεων ή και την ουσία των διαπραγματεύσεων. Ε, καλό θα ήταν να ακούσουμε και τις δύο πλευρές για τα θέματα αυτά. Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Και τώρα η Σκιώδης για δύο λεπτά. Ε, ο καθένας. Κολίν. Καρολίν. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε, ε, κυρία Κέρνικ. Ε, ευχαριστούμε για την, ε, τις παρατηρήσεις. Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμέναμε τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι χαιρόμαστε διότι υπάρχει διαφάνεια και η διαπραγματευτική εντολή δημοσιεύτηκε και ελπίζομαι ότι οι διαπραγματεύσεις θα προχωρήσουν ε, με διαφάνεια και θα μπορέσουμε να κάνουμε χρήσιμες ανταλλαγές απόψεων και να παρουσιάζουμε σωστά τα αποτελέσματα. Αυτό ελπίζω να συνεχιστεί και στο μέλλον. Κάποιες ερωτήσεις τώρα ή σχετικά με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Είπατε ότι συζητήθηκαν όλα τα κεφάλαια. Ερωτώ λοιπόν, τι γίνεται με την απελευθέρωση των υπηρεσιών, τι προσέγγιση επελέγει εδώ, ε, θετικός ή αρνητικός κατάλογος. Επίσης, ο γεωργικός τομέας, ξέρετε ότι εγκρίναμε ψήφισμα που λέει ότι τα ευαίσθητα προϊόντα θα πρέπει να ή να εξαιρεθούν από τις διαπραγματεύσεις. Σε ποιο βαθμό η Αυστραλία αντέδρασε σε αυτό, ε, τι πιστεύουν οι, οι διαπραγματευτές μας, οι εταίροι μας ε, για την ανάπτυξη. Πάντα μιλάμε για δυνατότητα ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, σε ποιο βαθμό προβλέπονται οι σχετικοί μηχανισμοί. Η Αυστραλία είναι και μέλος της ε, συνολικής και εταιρική σχέσης ε, για την ανταλλαγή προϊόντων. Το κεφάλαιο περιβάλλον παίζει ρόλο ε, εδώ και προβλέπονται και κυρώσεις προκειμένου περί παραβάσεων. Από πλευράς Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας δεν θα υπήρχε πρόβλημα λοιπόν. Τι λέει η ευρωπαϊκή πλευρά. Επίσης η καταπολέμηση της διαφθοράς. Έχει συμπεριληφθεί αυτό όπως και η φοροαποφυγή, η φοροδιαφυγή και είναι σημαντικό επίσης το θέμα της ισότητας των φύλων. Υπάρχει σχετικό κεφάλαιο, ποιες είναι οι διατάξεις και ε, συμπεριλαμβάνονται και γυναίκες στις διαδικασίες αυτές των ε, εμπορικών συμφωνιών και διαπραγματεύσεων που, θα, έχουν επιπτώσεις για τις γυναίκες. Ε, επίσης, ε, το... το ε, θέμα γενικότερα της περίθαλψης και των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος. Ευχαριστώ. Από το ECR, κύριε Μακλάρεν. Το ECR πάντα ήταν υπέρ των διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία και χαιρόμαστε που προχωράμε και προχωρούν διαπραγματεύσει αυτές και χαίρομαι για τη φιλοδοξία που επιδεικνύουν και οι δύο πλευρές στις συζητήσεις που γίνονται μέσα στις διάφορες ομάδες εργασίας που καλύπτουν πολλά θέματα σχετικά με την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει ε, αυτή την δέσμευση υπέρ των διαπραγματεύσεων, των εντατικών διαπραγματεύσεων και να εμείνουμε επίσης και στο χρονοδιάγραμμα που είναι αρκετά σφιχτό. Φυσικά και υπάρχει κάποια βεβαιότητα στην Αυστραλία. Και μετά από αυτά που είπε και ο κύριο Μόης, εγώ θέλω να ρωτήσω. Έχετε ε, πάρει τίποτα για την εντολή της Αυστραλίας όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις αυτές. Πάντως υπάρχει ένας νέος υπουργό εμπορίου, ίσως να έχετε επαφή μαζί τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι σε θέση να έχει αυτή την ελεύθερη πρόσβαση στις αγορές μέσα στους επόμενους μήνες. Και θα υπάρχει δυνατότητα για ειδικά κεφάλαια εμπορίου. Θα πρέπει να υπάρχουν ειδικές διατάξεις στο CTTP να προχωρήσουμε γρήγορα με τους κανόνες, ώστε να υπάρξει η κύρωση όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευχαριστούμε. Η Έλση Κατάινεν, Άλντε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πραγματικά και εγώ χαίρομαι που προχωρούν οι διαπραγματεύσεις και με την Αυστραλία και με τη Νέα Ζηλανδία. Οι χώρες αυτές είναι εμπορικοί εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι πεπισμένη που παρόλο που η παγκόσμια κατάσταση μπορεί να είναι δύσκολη, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια ολοκληρωμένη συμφωνία, οι περισσότερες χώρες θα αποφεληθούν. Ο κοινό στόχος για την Αυστραλία, την Νέα Ζηλανδία και την Ευρώπη είναι η συνέχεια στον ΠΟΕ έτσι ώστε να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο παγκόσμιο εμπόριο, εφόσον βέβαια υποστηρίζουμε κοινού κανόνες. Ακόμα και αν οι χώρες αυτές μοιάζουν πολύ, οι διαπραγματεύσει που κάνουμε τη μία και με την άλλη είναι ξεχωριστές, είναι πολύ διαφορετικές. Στη Γεωργία, για παράδειγμα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει ισορροπία στο τέλος Υπάρχουν λεπτοί τομεί ευαίσθητοι και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και τα συμφέροντα των Ευρωπαίων. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη της Επιτροπής από αυτού. Η Αυστραλία, η οικονομία της Αυστραλίας είναι μία από αυτές που αναπτύσσονται περισσότερο και είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική για την Ευρώπη. Αλλά και η Νέα Ζηλανδία βρίσκεται μπροστά από μας. Πάντως χαίρομαι για την προσπάθεια αυτή που γίνεται για μια συνολική διευθέτηση. Με την Νέα Ζηλανδία πρέπει να δούμε διάφορα διεθνή ζητήματα. Η προσέγγιση τους αντιστοιχεί σε αυτά που έχει τονίσει και σε προηγούμενες συμφωνίες της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, καταλαβαίνω ότι υπάρχει δυσκολία να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Ευχαριστούμε κύριος Μπούχνερ εκ μέρους των Πρασίνων, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η πρόθεση της νέας Αυστραλιανής κυβέρνησης ε, να αποχωρήσει από την κορυφή των Παρισίων ε, ανησυχεί και τους Αυστραλούς. Είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας άνθρακα η Αυστραλία. Από τις εκθέσεις του πρώτου γύρου βλέπω ότι η αμοιβαία πρακτική προκειμένου ε, ε, ε, συμφωνήθηκαν μελλοντικά μέτρα και έγινε ανταλλαγή πρακτικών προκειμένου περί συμφωνιών. Τι συγκεκριμένα έχει λεχθεί εδώ. Επίσης, αν όντως αποχωρήσει από τη Συμφωνία των Παρισίων η Αυστραλία, τι θα κάνει η Κομισιόν. Είναι αυτό κόκκινη γραμμή για μας στις διαπραγματεύσεις ή θα το δεχτούμε χωρίς άλλη κουβέντα. Νομίζω ότι ως μεγάλο εμπορικό μπλοκ στον κόσμο έχουμε κάποια ευθύνη που ξεπερνάει τα κέρδη και μόνο. Ε, ε, και σε αυτό ακριβώς θα ήθελα να παραπέμψω. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να υπενθυμίσω στην Επιτροπή ότι τον Ιούλιο στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου ενέκρινε ψήφισμα με ευρεία συνένεση όλων των πολιτικών ομάδων. Να μην υπάρχει εμπορική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών χωρίς να γίνεται μνήα στη συμφωνία των Παρισιών. Κουέ, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον πρέσβη και τον κύριο Μόιζε αλλά και τους σκιώδεις εισηγητές για τις προσπάθειές τους. Οι διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία προχωρούν αλλά τελικά πρόκειται περισσότερο για την αύξηση των μεταφορών προϊόντων από αυτές τις χώρες προς εμάς. Αυτό όμως δεν βλέπω πως συνάδει με τη Συμφωνία των Παρισίων. Στην Αυστραλία βέβαια και συμφωνούν, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το κόστο των μεταφορών. Πρέπει να λυθεί και αυτό υπόψη στην τιμή. Δεν είναι δυνατόν να φέρουμε προϊόντα από την άλλη άκρη του κόσμου και να κοστίζουν πιο φτηνά, σημαίνει ότι δεν λαβαίνουμε υπόψη μας το κόστος της μεταφοράς τους προς εμάς. Βρισκόμαστε στις δύο άκρες ε, του κόσμου και δεν είναι δυνατόν. Ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη πίεση εξαιτία ε, του εμπορίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε πρέπει να ξέρουμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις τι ακριβώς γίνεται λαμβάνεται υπόψη και αυτό το κόστος ή όχι. Τέλος, η ρυθμιστική συνεργασία, ρυθμίσεις, ε, κάτι που εμφανίζεται σαν είναι φιλικό προς τους καταναλωτές, τους εμπόρους κτλ. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει μόνο διάλογος για τις επιχειρήσεις και οι ευρωβουλευτές δεν έχουν καν πρόσβαση. Τελικά πρόκειται για μία τυποποίηση, δηλαδή από την πίσω πόρτα βάζουμε τις πολυεθνικές να διαπραγματεύονται εκείνες αντί για μας. Θέλω να ξέρω λοιπόν πώς ακριβώς γίνονται οι διαπραγματεύσεις, με ποια μορφή και να ξέρω κατά πόσο υπάρχουν πράγματι τέτοια δίκτυα διαπραγματεύσεων εκτός κοινοβουλίου. Ποιος επηρεάζει τελικά τις συμφωνίες αυτές στην πραγματικότητα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω κι εγώ να καλωσορίσω εδώ την κυρία Μινέρ που γύρισε από τις διακοπές. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Για την Αυστραλιακή είναι ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων μεταξύ της Αυστραλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει συζητηθεί ποτέ, είναι κάτι το οποίο έχει τεθεί. Υπάρχει πρόταση ρήτρα για ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ Ευρώπης και Αυστραλίας. Θα ήταν λογικό να το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όχι, χωρίς να υπάρχει αυτή η ρήτρα ελεύθερης κυκλοφορίας έχουν πρόσβαση στις αγορές. Άλλη ερώτηση, ή πρόταση τέλος πάντων, για τις προτάσεις ότι η Αυστραλία λέτε πρέπει να πληρώνει για την πρόσβασή της στην ευρωπαϊκή αγορά. Μα ακριβώ αυτό ζητάτε από το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα βάζει με το Ηνωμένο Βασίλειο έτσι κι αλλιώς εμείς δίνουμε 40 δισεκατομμύρια ευρώ, στερλίνες, αλλά εν πάση περιπτώσει πληρώνουμε εμεί λέτε, να πληρώνουμε για την πρόσβασή μα αγορές, αλλά η Αυστραλία όχι. Τώρα η έκθεση μετά τις πρώτες διαπραγματεύσεις. Εγώ δεν βρήκα και πολλά για τις διαπραγματεύσεις και τις προτάσεις όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα, που είναι ένα επίμαχο και ακαθόδες θέμα. στις εμπορικές συμφωνίες. Έπειτα για ενέργεια και πρώτες ύλες. Ποια είναι η θέση επ' αυτού. Το κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρει τα γεωργικά προϊόντα στο 19J, αλλά εγώ θα ήθελα κάποια στοιχεία που δεν υπάρχουν εδώ. Και τέλος, για την ουσία, το ιστορικό πλαίσιο, και έχει να κάνει εδώ και με τη χώρα μου, είναι ότι όταν εμείς οριστικά το 1975 μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε εκπνεύσει δηλαδή η η προηγούμενη συμφωνία. Εμείς είχαμε συμφωνία με την Αυστραλία, την οποία και καταργήσαμε. Και ο ορθολογισμός του να είναι κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι είναι πολύ πιο εύκολο, είναι πολύ πιο πιθανό να μπορεί κανείς να έχει εμπορικέ συμφωνίες. Λοιπόν, 40 χρόνια αργότερα εξακολουθούμε να συζητάμε για αυτά. Πάντως απαντήστε στην ερώτησή μου παρακαλώ για τη Γεωργία. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τον λόγο για αρκετά λεπτά στον πρέσβη της Αυστραλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την Επιτροπή σας και τους εισηγητές για τα σχόλια τα οποία έκαναν τη δική μας ε, πλευρά ήταν ο πρώτος γύρος ε, και επομένως τον περισσότερο χρόνο τον ε, δαπανίσαμε συζητώντας τον τρόπο και τη μεθοδολογία της διαπραγμάτευσης, το χρονοδιάγραμμα και βεβαίως ε, το πρόγραμμα ολοκλήρωσης ε, των διαπραγματεύσεων. Κατά την έννοια αυτή ε, θα συμφωνήσω με τα σχόλια που έκανε και η κυρία Κιόνικ σχετικά με το κλίμα και με το κατά πόσον ήταν πολύ θετική η συζήτηση. Κατά την άποψή μας είναι φιλόδοξη η διαδικασία. Ε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στην Αυστραλινή πλευρά πολλές ε, αμφιβολίες ε, και κάποια, κάποιες πιέσεις από την κοινή γνώμη και πραγματικά έπρεπε να γίνουν και κάποιες δηλώσεις σχετικά με ανοιχτό και δίκαιο εμπόριο. Ε, βεβαίως το χρονοδιάγραμμα θα είναι οπωσδήποτε φιλόδοξο και θα αποτελέσει πρόκληση και για τη μία και την άλλη πλευρά. Το ζήτημα είναι να βρεθούν λύσεις ε, στα προβλήματα τα οποία έχουν η μεν και η δε, αλλά να είναι και αμοιβαία αποδεκτές όσον αφορά τις ερωτήσεις σχετικά με την νέα κυβέρνηση, θα απαντήσω όσο πιο πολύ ε, μπορώ. με την νέα κυβέρνηση, ναι, ε, υπάρχει ε, ο Σένατορ Μπέρμιγχαμ, ο οποίος είναι ο νέος υπουργός που έχει αναλάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων και έχουμε και τον κύριο Μόρισον, ο οποίος όμως εξακολουθεί να έχει την θέση όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο, έτσι ώστε να υπάρχει και η σωστή συνέχεια μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Δεν έχω ακόμα δημοσιευμένο υλικό από πλευράς του γερουσιαστού Μπέρμπιγχαμ. Ε, ωστόσο, Νομίζω ότι ε, η Αυστραλινή κυβέρνηση είναι βέβαιο ότι θα παραμείνει ε, ε, προσιλωμένη στις αρχές της, των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τη Συμφωνία των Παρισίων, εξεπλάγει από την δήλωση ότι αποφασίστηκε η απόσυρση της Αυστραλίας από την Συμφωνία των Παρισίων. Ε, η Αυστραλία έχει αναλάβει δεσμεύσεις ε, όσον αφορά το πλαίσιο ε, της Συμφωνίας των Παρισίων και βεβαίως ε, είμαστε προσιλωμένοι στο να βρούμε λύσεις όσον αφορά αυτές τις μεγάλες ε, προκλήσεις. Η θέση μας είναι ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα χρονικά όρια εντός των οποίων πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και φρονούμε ότι οπωσδήποτε αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κυρίως η ποιότητα την οποία δεν προτιθέμεθα θα να θυσιάσουμε υπέρ της ε, ταχύτητος. Το θέμα δεν είναι να γίνουν τα πράγματα γρήγορα, αλλά να γίνουν σωστά. Ε, και πιστεύω ότι ε, όλα θα πάνε καλά όσον αφορά την γεωργία. Όπως έχω ήδη ε, ξαναπεί, αυτό που προσπαθούμε είναι να επιτύχουμε μια συνολική συμφωνία, comprehensive deal, ε, όχι εξαιρέσεις προϊόντων και ε, ζητημάτων από το θεματολόγιο. Δεν θέλουμε τέτοιες αποκλήσεις και αποκλισμούς. Ενδεχομένως καλύτερα το πακέτο είναι να είναι μικρότερο αλλά να είναι πιο συνεκτικό και βεβαίως θέλουμε όσο γίνεται περισσότερα αποτελέσματα. Για τις ε, υπηρεσίες ε, ε, θέλουμε το θέμα των λιμενικών, των υπηρεσιών λιμένων ε, και το θέμα ε, της δημιουργίας ενός καλού περιβάλλοντος για την υποδοχή των εταιριών και από τη μία και από την άλλη πλευρά να είναι σε σωστά επίπεδα. Θέλουμε διατάξεις οι οποίες θα δεσμεύουν τις κυβερνήσεις και από τις δύο πλευρές και κάποια τελικά σχόλια σε σχέση με με τις ε, διμερείς ε, προσπάθειες. Ε, να σας πω ότι από τη δική μας πλευρά εμείς προσπαθούμε να κινηθούμε σωστά και όσον αφορά τον παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίων. Εμείς ε, θέλουμε ε, να προωθηθούν και τα θέματα των πολυμερών ε, συμφωνιών αλλά και το θέμα του Δικαστηρίου Επίλυσης των Επιχειρηματικών Διαφοριών. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κιόνιχ. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τα ερωτήματα τα οποία θέσατε. Θα ξεκινήσω από τις πρώτες ερωτήσεις, γιατί έπρεπε να ξεχωριστούν ε, οι διαπραγματεύσεις ε, για την Αυστραλία και για την ε, Νέα Ζηλανδία. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο με την έννοια ότι μιλάμε για δύο διαφορετικές χώρες, δύο διαφορετικές οικονομίες, ενδεχομένως με διαφορετικές προτεραιότητες και από πλευράς Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, αλλά και από, τις, από τη δική μας πλευρά αποφασίσαμε να μην κάνουμε κοινέ διαπραγματεύσει, αλλά η απόφαση αυτή ελήφθη πριν από πολύ καιρό. Είμαι επεπισμένη ότι αυτό είναι ο σωστός τρόπος ε, για να προχωρήσουμε και ευελπιστούμε ότι θα ε, καταφέρουμε να έχουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ε, προόδου και στις δύο διαπραγματεύσεις. Ο κύριος Πρέσβης προηγουμένως αναφέρθηκε στο θέμα αυτό και είπε ότι και εκείνος ελπίζει γρήγορη πρόθεση των διαπραγματεύσεων. Βεβαίως δεν έχουμε και πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ε, απ' την άλλη πλευρά είναι γεγονός ότι και το θέμα των ε, εντολών πήρε περισσότερο χρόνο από ό,τι ε, ελπίζαμε. Ούτως ή άλλως, ανάμεσα από το πρώτο και το δεύτερο γύρο πάντα θα υπάρχει, θα συνεχίζεται η εργασία. Ξεκινήσαμε αργά πάντως και είναι γεγονός ότι υπάρχουν άλλα ζητήματα τα οποία προκύπτουν και παίρνουν σειρά κατά κάποιο τρόπο, οπότε θα, είναι, θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα όσον αφορά τις διαβουλεύσεις, ε, τις επιγραμμικές διαβουλεύσεις online consultations. Χρειάζεται χρόνος για να δούμε και τις απαντήσεις. Κάποιες από τις επιχειρήσεις ή τις ε, ε, οργανώσεις ζήτησαν να μην προωθηθούν οι πληροφορίες που έδωσαν. Πέρα από αυτό όμως, εμείς είμαστε αρκετά ανοιχτοί στη δημοσιοποίηση και το πιο πιθανό είναι να υπάρχει μια compilation των απαντήσεων. Πάντως, οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο ε, μπορούμε ε, ωραιότατα να ε, βάλουμε στο διαδίκτυο. Τώρα, το κείμενο υπευλήθη αρκετά αργά και οι δύο πλευρές πρέπει ε, να προχωρήσουν με τις συνήθεις τους προβλεπόμενες διαδικασίες και επομένως ε, είναι νωρίς για να μιλάμε για λύσεις. Ε, οπωσδήποτε η κάθε πλευρά έχει κάποιες δυνατές λύσεις κατά νου θα τις ελέγξουμε και θα τις συζητήσουμε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Όσον αφορά την πρώτη ανταλλαγή προσφορών, βεβαίως ξεκινήσαμε τη συζήτηση επί των παραμέτρων της προσφοράς. Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε την πρώτη ανταλλαγή προσφορών τον Νοέμβριο. Προσπαθούμε να κρατήσουμε έτσι κάποια παράλληλη ε, δράση με τα διάφορα κεφάλαια των ε, ε, διαπραγματεύσεων ε, η επικεφαλής ε, διαπραγματεύτη όταν θα είναι εδώ το Σεπτέμβρη θα το συζητήσει, θα έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή να το συζητήσουμε μαζί της. Ε, αυτό που θέλουμε εμείς, όπως είπα και προηγουμένως, είναι οι γεωγραφικές ενδείξεις από την πλευρά της Αυστραλίας η πρόσβαση στη γεωργική αγορά κατά την άποψή μας θα πρέπει να προχωρήσουμε κάπως παράλληλα, όχι ακριβώς παράλληλα, αλλά να γίνει μια προσπάθεια παρόλα αυτά. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν κάποια παράλληλη δράση όσον αφορά την αντιμετώπιση των κεφαλαίων όσον αφορά τον διάλογο εμπορικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια είναι συνήθις και διαρκής με την Αυστραλία και με την Νέα Ζηλανδία προσπαθούμε να μην ε, μπαίνουμε ε, ε, πολύ σε ζητήματα τα οποία συζητούνται στα πλαίσια της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου. Υπάρχουν βέβαια και τα ζητήματα τα οποία αφορούν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και τα οποία συζητιούνται. Επίσης, συνήθως έχουμε μια καλή συζήτηση σε σχέση με το τι συμβαίνει και στις άλλες διαπραγματεύσεις γιατί και αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον. Επομένως, προς ώρα συνεχίζουμε την προσπάθεια που ξεκινήσαμε ε, και θα γίνεται και ε, άπαξ άπαξιότητας μια συνάντηση ε, κατά παράλληλο τρόπο. Όσον αφορά τις υπηρεσίες και το, το κείμενο δεν έχει υποβληθεί ακόμα δεν θα αποφασίσουμε μόνο για την αρχιτεκτονική, μάλλον δεν έχουμε αποφασίσει πλήρως την αρχιτεκτονική, τη δομή του κεφαλαίου ε, για τις υπηρεσίες. Ε, έχουμε το δε θέμα του negative listing ε, όσον αφορά τις υπηρεσίες, αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν έχουν ληφθεί ακόμα αποφάσεις. Από την άλλη πλευρά, έχουμε πολλά κοινά και κοινή αντιμετώπιση σε άλλα ζητήματα. Επομένως, ε, για τις υπηρεσίες ε, υπάρχει κοινή κατανόηση, υπάρχουν πολλά πεδία τα οποία συμμεριζόμαστε. Ε, όσον αφορά τις παραμέτρους για τις προσφορές υπηρεσιών στον επόμενο γύρο, περιμένουμε να είμαστε πιο έτοιμοι, αλλά θα ξανασυζητηθεί αυτό από, τους επικεφαλείς διαπραγματευτές. Όσον αφορά τα TST, και από την ε, έκθεση ε, θα έχετε δει ότι έχουμε υποβάλει ο καθένας ε, τις απόψεις του. Έχουμε επίσης ένα σχέδιο δράσης 15 ε, θεμάτων, σημείων για την καλύτερη υλοποίηση των ε, όσων σχετίζονται με τα TST. και μέσω αυτών των 15 σημείων ευελπιστούμε ότι θα ε, βελτιωθούν τα πράγματα όσον αφορά τη Συμφωνία των Παρισίων. Παρατηρήσεις εκτός μικροφώνου από την κυρία Αρενά δεν ακούν οι διερμηνείς όσον αφορά την ε, Συμφωνία των Παρισίων. Πιστεύω ότι ακούσαμε από την πλευρά του πρέσβεως τα ε, σημαντικά και οπωσδήποτε υπάρχει ε, ε αναμφίβολα ε, σεβασμός ε, της συμφωνία των Παρισίων. Θα δούμε πώς θα παρουσιαστεί αυτό και στο κείμενο. Σχετικά με τη διαφθορά, κεφάλαιο για τη διαφθορά. Έχουμε διατάξεις ε, για την ε, διαφθορά. Τις είχαμε αναφέρει στη Συμφωνία για το Μεξικό και μετά στη Συμφωνία με τη Χιλή. Έχουμε επίσης ε, τάξεις οι οποίες αφορούν την ισότητα των φύλων όμως για την πλευρά, για την συμφωνία με την Αυστραλία δεν προτιθέμεθα προς ώρας να υποβάλλουμε τέτοια διάταξη, δηλαδή που θα αφορά είτε την διαφθορά είτε την ισότητα των φύλων. Πρόθεσή μας για προσόραση είναι να μην γίνει τέτοια αναφορά στα κείμενα. Όσον αφορά το ε, ψηφιακό εμπόριο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για, το, αντιμετώπιση του ψηφιακού ε, ε, ε ηλεκτρονικού εμπορίου. Στον επόμενο γύρο θα αναφερθούμε σε αυτά. Είναι πάντως ε, σαφές ότι οπωσδήποτε θα υπάρξουν κάποιες διατάξεις όσον αφορά τα θέματα αυτά. Όπως είπα και προηγουμένως έχουμε διαφορετική προσέγγιση ε, για τα θέματα αυτά μεταξύ Αυστραλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ε, όσον αφορά τώρα τις ξεχωριστές ε, διαπραγματεύσεις, κάτι υπόθηκε το οποίο μου διέφυγε. Υπάρχουν μηχανισμοί πάντως ε, και για τα SIA και για τις διαπραγματεύσεις. Πάντως θέλουμε πάντα και συχνά την γνώμη της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά και αυτές τις διαπραγματεύσεις αλλά και άλλες διαπραγματεύσεις. Όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία, όχι, δεν υπάρχει καμία ρήτρα συγκεκριμένη και ρητή όσον αφορά την ελεύθερη ε, κυκλοφορία. Ε, υπάρχει κάποια αναφορά ε, όσον αφορά τις επενδύσεις και είναι με και τους επιχειρηματίες και τη δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας τους αλλά είναι μια τυπική ε, αναφορά που γίνεται και σε άλλες συμφωνίες και οπωσδήποτε δεν είναι συγκεκριμένη η Συμφωνία Ελεύθερης ε, Κυκλοφορίας. Όσον αφορά ε, τα γεωργικά προϊόντα, δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοούσατε. Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στην πρόσβαση στην αγορά. Όπως είπα και προηγουμένως, το θέμα αυτό ε, θα το αναλύσουμε όταν θα έχουμε την πρώτη, ανταλλαγή, συγγνώμη, την πρώτη ανάλυση των προσφορών. Όσον αφορά τις πρώτες ύλες, και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, όσον αφορά τη συμφωνία με την Αυστραλία, είναι από τα πιο πρόσφατα ε, κεφάλαια ε, στι ε, διαπραγματεύσει. Μερικέ φορέ έχουμε διατάξει, μερικέ φορές προβίσει, μερικέ φορές έχουμε κεφάλαια, chapters. Οπωσδήποτε η Αυστραλία είναι σημαντικό πάροχο πρώτων και προμηθευτή μάλλον πρώτων υλών. Επομένω μα ενδιαφέρει το θέμα και είναι σημαντικό να έχουμε κοινέ απόψει έτσι ώστε να παραμείνουν ανοιχτέ οι αγορέ. Πάντως όπως είπα και προηγουμένως Μόλι ξεκίνησαν αυτέ οι συζητήσει, επομένω όλα αυτά παραμένουν ανοιχτά. Δεν νομίζω να έχω τίποτα άλλο να Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Συμπέρασμα. Ο εισηγητή μα. Ωραία. Τι μου μένει εμένα από όλη αυτή τη συζήτηση είναι ότι γενικά υπάρχει στήριξη από την Επιτροπή μας, βέβαια με κάποιες αποχρώσεις που έχω σημειώσει και θα προσπαθήσω να τις συμπεριλάβω στο τελικό μου κείμενο. Θέλουμε μια στέρεα συνολική συμφωνία. Ε, κοιτάμε πρώτα την ποιότητα και μετά την ταχύτητα Θέλουμε βέβαια σε αυτή τη θητεία της Επιτροπής να τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις και βέβαια να προλάβει να ψηφίσει και αυτό το Κοινοβούλιο. Και το Παρίσι, ναι, να ληφθεί υπόψη. Ακούσαμε και τον πρέσβη της Αυστραλίας ότι φυσικά και θα τηρήσει αυτές τις δεσμεύσεις. Και εννοείται ότι για τα θέματα αρχής ε, φυσικά και δεσμευόμαστε υπέρ της Συμφωνίας των Παρισιών. Τώρα πώς αυτό θα αντικατοπτρίζεται μέσα στο κείμενο δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή. Πάντως είμαι αρκετά αισιόδοξο για το μέλλον. Καλώς. Ευχαριστούμε. Σημείο 15 τώρα. Κάτι παρόμοιο για τη Ζηλανδία αυτή τη φορά. Λοιπόν, για πείτε μας τι γίνεται στις διαπραγματεύσεις με τη Νέα Ζηλανδία, κυρία Γκρίζουν. Ωραία. Λοιπόν, ο γύρος με την Νέα Ζηλανδία έλαβε χώρα λίγες εβδομάδες μετά από εκείνον με την Αυστραλία, στις Βρυξέλλες επίσης. Υπάρχουν οι προτάσεις, τις έχουμε υποβάλει και τις έχουμε στείλει και στην Επιτροπή σας. Η διαπραγμάτευση αυτή συζητάει όλα τα κεφάλαια, τα εμπορικά, όπου οι διαπραγματεύτες από πλευράς Νέας Ζηλανδίας ήταν διαθέσιμοι. Όπως γίνεται και με την Αυστραλία, έτσι και εδώ είδαμε ότι οι διαπραγματευτές από πλευράς Νέας Ζηλανδίας ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι, καλοί επαγγελματίες. Είχαμε ένα πολύ καλό σημείο κίνησης. Έγιναν και λεπτομερείς συζητήσεις, ακριβώς γιατί ήταν δύο εβδομάδες μετά την Αυστραλία, οπότε η Νέα Ζηλανδία είχε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή της να προετοιμαστεί κατά κάποιο τρόπο σχετικά με τις δικές μας 12 προτάσεις και διάφορα άρθρα συμφωνήθηκαν ήδη, όπως βλέπετε και στα πρακτικά. Επίσης προσπαθήσαμε να βρούμε και λύσεις στην ε, διατύπωση. Αν δεν έχουμε ακριβώς το ίδιο κείμενο, τουλάχιστον υπάρχει μια σύγκληση. Όπως και με την Αυστραλία, έτσι και εδώ, υπήρξε μεγάλη συνοχή για πάρα πολλά κεφάλαια και δεν μας ε, εκπλήσει αυτό δεδομένου του διευρυμένου πεδίου εφαρμογή. Ξέρουμε πολύ καλά πάντως πού θα είναι οι δυσκολίες. Γεωργία, δηλαδή γαλακτοκομικά, πρόβιο, ε, ονομασίες προέλευσης, γεωγραφικές ενδείξεις. Ξέρουμε λοιπόν πού θα είναι τα εμπόδια μπροστά μας και εκεί θα επικεντρωθούμε για να βρούμε λύσεις. Πάντως ήταν θετικό το κλίμα. Θα συνεχιστούν οι συζητήσεις τώρα το φθινόπωρο. Τον Οκτώβριο θα έχουμε τον πρώτο γύρο στη Νέα Ζηλανδία, που θα είναι ο δεύτερος συνολικά. Και θα υποβάλουμε κάποιες νέες προτάσεις διατύπωσης κυρίως για τη διαφάνεια, καλές ρυθμιστικές πρακτικές, βιώσιμη ανάπτυξη, υπηρεσίες και SPS. Για όλα αυτά λοιπόν είμαστε σε καλό δρόμο, έχουν μπει στο αυλάκι. Κάπως πιο γρήγορα από ό,τι έγινε με την Αυστραλία. Αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ε, διάφορες διαπραγματεύσεις. Δεν είναι ότι θα πάμε πιο γρήγορα με την Νέα Ζηλανδία από ότι με την Αυστραλία. Ε, απλώς και στην περίπτωση Αυστραλίας και στην περίπτωση της Νέας Ζηλανδίας θέλαμε έτσι καλλιώς να πάμε γρήγορα. Ε, κρατάμε όμως παραπάνω από ό,τι με άλλους ε, εταίρους. Σωστά, ο κύριος Κάσπαρη. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, και αυτό το καλοκαίρι είδαμε ότι δεν σταθεροποιήθηκε η διεθνής κατάσταση και μετά από πολλά χρόνια προσπαθούμε να βάλουμε σε νέα βάση τις εμπορικές μας σχέσεις και με τη Νέα Ζηλανδία και να το τεκμηριώσουμε αυτό. Υπάρχει η ευκαιρία. Τώρα αποσύρονται όλο και περισσότερο οι ΙΠΑ από την περιοχή, η Κίνα παρουσιάζεται με αυξημένη αυτοπεποίθηση στην ίδια αυτή περιοχή και οι εμπορικές μας σχέσεις με την ε, Νέα Ζηλανδία μπορούν να σταθεροποιηθούν μέσα από μια καινούργια συμφωνία. Επίσης έχουμε μια τεράστια ε, ε, ευκαιρία λόγω της μειωμένης επιρροής των ΙΠΑ και της αυξημένης επιρροής άλλων εταίρων να δούμε κάποια θέματα εκ νέου ε, που αφορούν τα πρότυπα, την ασφάλεια, όλα αυτά να κατοχυρωθούν στην συμφωνία και ελπίζομαι ότι θα μπορέσουν ε, διεθνώς να ρυθμιστούν. Οι διαπραγματεύσεις προετοιμάστηκαν καλά. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, εμείς ζητήσαμε την έγκαιρη έναρξη των διαπραγματεύσεων. Διατυπώνουμε σαφώς στο ψήφισμα ότι υπάρχουν προϋποθέσεις και όροι που θεωρούμε σημαντικούς για τα πρότυπα, για, για την, ε, τις υπηρεσίες ε, γενικού ενδιαφέροντος ε, σε περιφερειακή βάση και αυτά ήταν θέματα που ίσχυσαν και στη διαπραγματεύση με τον Καναδά. Ελπίζω να προχωρήσουμε γρήγορα οι διαπραγματεύσεις κυρία Κόνικ, το ταχύτερο δυνατό να τελειώσουμε για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Επίσης, καλό είναι οι επιχειρήσεις μας να έχουν ε, όσο γίνεται πιο γρήγορα τις βελτιωμένες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά της Νέας Ζηλανδίας και ε, επίση ε, καλό είναι να δείξουμε και σε άλλους εμπορικούς εταίρους πώς μπορεί να διαμορφωθεί μια σωστή συμφωνία, πώς μπορούν οι διεθνείς εμπορικές σχέσεις να διατηρούνται και έτσι να βελτιώνεται και να σταθεροποιείται η κατάσταση γενικότερα για τον, τους πολίτες μας. Ε, καλό είναι να μας στείλετε, όπως είπατε, έγκαιρα τα σχετικά έγγραφα και να δείτε πώς θα ενημερώσετε επαρκώς ε, τον, τους ενδιαφερόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη συμφωνία με την Νέα Ζηλανδία και να υπάρχει διαρκής ενημέρωση για να αποφεύγονται ενδεχομένως σφάλματα. Ναι, βεβαίως νομίζω ότι σε όλους τους εμπορικούς εταίρους πρέπει να σταλεί αυτό το μήνυμα. Και τώρα η Σκιώδης, η Καρολίνα είναι η πρώτη. Ευχαριστώ. Θέλω να καλωσορίσω και εγώ τον πρέσβη. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Ακούσαμε πολλά για την Αυστραλία, πολλά τα ίδια ισχύουν πολύ και για τη Νέα Ζηλανδία. Ε, μιλάμε για ταχύτητα, ε, αλλά πάνω απ' όλα για ποιότητα. Ε, θα πρέπει να πάρει το χρόνο που χρειάζεται η διαπραγμάτευση, ούτως ώστε το αποτέλεσμα να είναι καλό και να μπορούμε να το υποστηρίξουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία ερώτηση για τις βασικές συμφωνίες του ΟΗΕ. Θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς ε, ε, διαδικασίες ακολουθούνται. Πριν από το τέλος των διαπραγματεύσεων πρέπει να γίνει επικύρωση και εφαρμογή τους. Ε, δεν νομίζω αν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις θα έχουμε πρόβλημα με την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία. Ε, η Νέα Ζηλανδία πώς ε, αντιδρά σε σχέση με τις ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει προσέγγιση στη θέση σχετικά με τα διάφορα προϊόντα. Επίσης η Νέα Ζηλανδία τι διαδικασίες ακολουθεί για το ψηφιακό εμπόριο, το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ζούμε σε παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Η μεταφορά δεδομένων, η ροή δεδομένων είναι σημαντική. Τι συγκεκριμένες προτάσεις, αν υπάρχουν σε αυτό το στάδιο, έχουν γίνει. κύριε Ευχαριστώ για την ε, Νέα Ζηλανδία. Τις ίδιες ερωτήσεις που έκανα και πριν για την πρόσβαση στα αγαθά, τις ε, συνθήκες του εμπορίου. Απαντήσατε βέβαια στην προηγούμενη περίπτωση. Πάντως στις διαπραγματεύσεις προσπαθούμε να έχουμε κάποια ισορροπία με την Αυστραλία, αλλά υπάρχει περίπτωση να επιταχυνθεί κάπως περισσότερο η διαδικασία με την Νέα δηλαδή περισσότερο από ό,τι με την Αυστραλία. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα με τον ένα τέρο να επιταχύνουμε περισσότερο εφόσον το επιθυμεί από ό,τι με τον άλλον. Ο Κλάους Μπούχνερ για τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ. Επανέρχομαι στο θέμα της διευθέτησης των διαφορών. Υπάρχουν προτα... Υπάρχει πρόταση. Ποια είναι ακριβώς και πού βρίσκονται τα βασικά προβλήματα από, από, την πλευρά της Νέας Ζηλανδίας. Επίσης, αναφέρθηκε το κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, εδώ βλέπουμε να συμπλέουν οι δύο πλευρές. Τι θέλουμε όμως, θέλουμε ένα εφαρμόσιμο κεφάλαιο με μηχανισμό κυρώσεων ή όπως λειτουργούσε μέχρι τώρα, όπου περιοριζόμαστε σε ωραία μεγάλα λόγια. Δηλαδή θα ε, πρέπει να έχουμε και τη δυνατότητα εφαρμογής. Η κυρία Μινέρου. Ευχαριστώ. Όπως και με την Αυστραλία, έτσι και με τη Νέα Ζηλανδία, τα ίδια θέλω να ρωτήσω και δεν πήρα καν απάντηση σε αυτό που ρώτησα για την Αυστραλία, οπότε θα το ξαναρωτήσω. Λαμβάνετε υπόψη το κόστος μεταφοράς στην τιμή στις διαπραγματεύσεις αυτές. Δεύτερον, πώς ε, ασχολούμαστε ακριβώς με τις διαπραγματεύσεις και υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες που κάνουν διαπραγματεύσεις εκτός κοινοβουλίου. Ποιες είναι αυτές, θα ήθελα να το ξέρω. Τι δίκτυα υπάρχουν δηλαδή εκτός από τις επίσημες. David Μάρτιν. Ευχαριστώ. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε τις νέες ε, ρήτρες διασφάλισης όσον αφορά τη Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία και το Βιετνάμ, τις σχετικές συμφωνίες. Οπότε εδώ σε αυτή την περίπτωση θα συμπεριλάβουμε και την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Θα προκαταβάλουμε δηλαδή τα πράγματα για να συμπεριλάβουμε και αυτές τις δύο χώρες. Τώρα για τα σχόλια της ΕΜΑ και του συγητή για την ταχύτητα. Ωραία, καλή ταχύτητα, αλλά δεδομένου ότι έχει τους καλύτερους διαπραγματευτές στον κόσμο, Νέα δηλαδή εκτός φυσικά από τους δικούς μας εννοείται, έχει οικονομία που ενδιαφέρεται για την κοινωνία, το περιβάλλον έχει καλές ε, προδιαγραφές δεν βλέπω για ποιο λόγο να μην προχωρήσουμε με ταχύτητα και να ολοκληρώσουμε αυτή τη συμφωνία γρήγορα, ώστε να αποτελέσει και ένα καλό παράδειγμα. Η φήμη μα είναι συνήθως ότι καθυστερούμε στις διαπραγματεύσεις αυτές, οπότε μήπως είναι μια καλή ευκαιρία να ανατρέψουμε αυτή τη φήμη την κακή που έχουμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντάτσμορθ. Δεν ξέρω αν είδατε το έργο Groundhog Day όπου ο ήρωας την ίδια μέρα ξανά και ξανά επαναλαμβάνεται. Αυτό λοιπόν γίνεται εδώ τώρα νομίζω. Οι ερωτήσεις μου είναι ακριβώς οι ίδιες όπως αυτές που είχα για την περίπτωση της Αυστραλίας. Όμως, πιο συγκεκριμένα, όπως γνωρίζει εκπρόσωπος της Επιτροπής, αλλά όχι και όλοι οι συνάδελφοι, η γεωργία είναι πολύ πιο σημαντική για την οικονομία της Νέας Ζηλανδίας από ό,τι για της Αυστραλίας. Και εδώ δεν υπάρχει περίπου τίποτα για τη Γεωργία. Το ψήφισμα προτείνει το κοινοβουλευτικό, έτσι, ότι θα πρέπει να υπάρχουν ποσοστώσεις και να υπάρξουν και μεταβατικές περίοδοι. Το στηρίζει αυτό η Επιτροπή, αυτό κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα τι γίνεται με το κεφάλαιο που αφορά τη γεωργία, θέλω να ξέρω. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Πρέσβης της Νέας Ζηλανδίας τώρα, παρακαλώ να αντιδράσει. Ο κύριος David Βέλλαντ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά που ξαναβρίσκομαι εδώ πάλι. Ευχαριστώ και εσάς και τα μέλη της Επιτροπής για το ενδιαφέρον και ημών και του Κοινοβουλίου συνολικότερα για τη Νέα Ζηλανδία. Ε, είμαστε υπέρ της συνεργασίας ε, στενότερης, διαφανέστερης και όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις βεβαίως ε, θα πρέπει να συμφωνήσει με αυτήν και το Κοινοβούλιο. Ε, εμείς όπως γνωρίζετε έχουμε παλιές και ισχυρές ε, σχέσεις που έγιναν πιο βαθιές σύν το χρόνο. Ε, μαζί δίνουμε μάχες στα διεθνή φόρα για να με διεθνή προβλήματα. Η κυρία Μογκυρίνη ήταν στο Wellington τελευταία, είπε ότι δεν είναι πολλές οι χώρες που έχουν την ιστορία της Νέας Ζηλανδίας ε, με την, ε, σε σχέσεις με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Το CFTA είναι μεγάλη προτεραιότητα συμφωνία και είναι ένα μήνυμα της δέσμευσης υπέρ της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Θα θυμάστε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση πίεσε για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και η νέα ε, κυβέρνηση συνασπισμού προχώρησε στεναρά με τις διαπραγματεύσεις και οι τα δύο μέρη ε, προχώρησαν πολύ κατά τη διάρκεια των πρόσφατων επισκέψεων. Εμείς ε, πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι η διερευνητική διαδικασία με την Κομισιόν προχώρησε πάρα πολύ καλά, όπως προαναφέρθηκε. Ε, η κυρία Κόνικ περιέγραψε με ακρίβεια την κατάσταση. Πιστεύουμε ότι είναι υψηλή πολιτική δέσμευση και θέλουμε ένα υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα το ταχύτερο δυνατόν από τη διαπραγμάτευση. Ε, ε, θέλουμε, έχουμε υψηλά πρότυπα και για το εμπόριο και για μια ε, εμπορική πολιτική χωρίς αποκλεισμούς, ποιότητα και ταχύτητα. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κινηθούμε γρήγορα, όχι όμως σε βάρος μιας καλής ποιότητας συνολικής συμφωνίας. Είμαστε πολύ φιλόδοξοι για το αποτέλεσμα ε, Ελπίζουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι φιλόδοξη. Ε, η Νέα Ζηλανδία έχει πρόσφατα ε, ακολουθήσει, εγκρίνει εμπορική πολιτική στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βοηθήσει τις γυναίκες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την αλλαγή του κλίματος, περιβαλλοντικά θέματα, την εργασία, την ισότητα των φύλων και άλλα. Το, ε, επίσης ε, για τη διαφάνεια όπως είπα ε, θα συνεχίσουμε να έχουμε ανοιχτό το κανάλι επικοινωνίας με το Κοινοβούλιο. Πολλοί αναφέρθηκαν στην Γεωργία με λεπτομέρειες. Εμείς θέλουμε μεγάλη κάλυψη του τομέα αυτού στην ε, συμφωνία γιατί είμαστε σε μειονεκτική θέση σε σχέση με την Ευρώπη στο παρελθόν και θέλουμε ε, ισότιμους όρους. Πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν να υπάρξει συνολική συμφωνία χρησιμοποιώντας κάποια από τα εργαλεία που αναφέρθηκαν χωρίς την εξαίρεση προϊόντων. Πιστεύουμε ότι οι διαπραγματεύσεις ε, μπορούν να εξαλείψουν αυτές τις διαφορές έτσι όπως εξελίσσονται. Τώρα, για τις υπηρεσίες περιμένουμε να δούμε το κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά. Εμείς ε, στηριζόμεθα στο κείμενο της Ευρωπαϊκής, στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούμε να συνεργαστούμε. Βέβαια και σε κάποιους τομείς θα υποβάλλουμε τις δικές μας ιδέες. Αλλά έχουμε ως βάση το κείμενό σας. Θα δούμε τι θα γίνει με τις υπηρεσίες Υπάρχουν και κάποια νέα θέματα που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το ψηφιακό εμπόριο είμαστε, ε, τελειώσαμε τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων. Ε, νομίζω ότι ε, μπορούμε και την ιδιωτικότητα να την προστατεύσουμε, αλλά και την καλύτερη συνεργασία. Έχουν γίνει πολλά. Έχουμε συμφωνήσει για πολλές διατάξεις ε, στο, στα κεφάλαια και ε, έχουμε εξετάσει και το θέμα της διαδικασίας διαμεσολάβησης. Αυτό είναι καινούριο θέμα και κοιτάμε τις προτάσεις της Επιτροπής. Ξέχασα το θέμα του Διεθνούς ε, Οργανισμού Εργασίας. Έχουμε κυρώσει 6 από τις 8 συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου ε, μπορούμε να δεσμευτούμε υπέρ των ε, αρχών που αναφέρονται εκεί. Υπήρχε κάποιο θέμα ερμηνείας δύο από το ε, συμβάσεις του ΔΟΕ, αλλά μπορώ να σας βεβαιώσω ότι παρακολουθούμε τους στόχους των και τις διατάξεις και συμφωνούμε με αυτές. Και για να ολοκληρώσω, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να σας μιλήσω τα πράγματα προχωρούν καλά. Προσβλέπω στον επόμενο γύρο στο Wellington τον Οκτώβριο και την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε μια καλή συμφωνία. Ευχαριστώ. Η κυρία Κιόνιχ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω με την πιο δημοφιλή ερώτηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Όταν μιλάμε για ε, χρόνου έναντι ποιότητος, ε, νομίζω ότι όλοι έχουμε δίκιο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε όσο γίνεται γρηγορότερα με τις διαπραγματεύσεις με τη Νέα Ζηλανδία, αλλά αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι θα θυσιάσουμε ε, την ε, ποιότητα. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό και από τις δύο πλευρές, αλλά νομίζω ότι ταυτόχρονα αποτελεί κοινό στόχο η γρήγορη προώθηση ε, των εργασιών. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρξουν διαβουλεύσεις, θα πρέπει να εξευρεθούν λύσεις μεταξύ των διαφόρων διαπραγματευτικών γύρων. Θα πάμε και στην Νέα Ζηλανδία σύντομα, στον Οκτώβρη και μετά θα αποφασίσουμε πού και και πότε θα γίνει ο επόμενος γύρος. Είπαμε ε, πάντως ότι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ε, και εργασία μεταξύ των διαφόρων ε, γύρων αν πρόκειται αυτό να βοηθήσει να προχωρήσουμε. Είναι, υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά αλλά υπάρχει και κοινή διάθεση για το είναι γεωργία αλλά υπάρχει διάθεση να βρεθούν λύσεις ε, απελευθέρωση η πλήρηση όχι καθώς επίσης ε, και πρόσβαση στην αγορά ε, αυτά είναι τα ζητήματα τα πιο κεντρικά τώρα όσον αφορά συγκεκριμένε λύσεις θα πρέπει να περιμένουμε θα πρέπει να ελέγξουμε τις προσφορές για την πρόσβαση στην αγορά και μετά θα δούμε είμαστε πάντως υπέρ ανοιχτής πρόσβασης, αλλά θα πρέπει να δούμε ε, ε, επιτάπητος να θέσουμε όλοι τις ε, προσφορές οι διαπραγματεύσει μπορεί να περιλαμβάνουν παρόμοια στοιχεία, αλλά διαφέρουν ε, η καθεμία από την άλλη. Πάντως, με την ε, συμφωνία αυτή ε, θέλουμε να δείξουμε ότι όχι μόνο συμφωνούμε με τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου FTA, αλλά προσπαθούμε να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο το θεματολόγιο των των ε, ε, συμφωνιών και των διαπραγματεύσεων. Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή, ε, πριν από τον πρώτο γύρο. Θα δούμε ποιε θα είναι οι προτάσεις οι οποίες θα προκύψουν από πλευρά ε, της Νέας ε, Ζηλανδίας και να δούμε εάν και κατά πόσον μπορούμε να ε, συμφωνήσουμε. Οπωσδήποτε μας ενδιαφέρει να προωθήσουμε σε μια χώρα όπως, όπως η Νέα Ζηλανδία μια προοδευτική, ένα προοδευτικό θεματολόγιο όσον αφορά ψηφιακό εμπόριο ε, και γενικότερα όσον αφορά ε, τις υπηρεσίες. Όπως είπε και ο κύριος Πρέσβης, δεν έχουμε ακόμα κείμενο, αλλά για το ψηφιακό εμπόριο μπορώ ήδη να πω ότι η Κομισιόν έχει βάλει ε, στο διαδίκτυο ένα γενικό σχόλιο που αφορά ακριβώς το θέμα αυτό. Η εργασία όμως συνεχίζεται. σχετικά με την επίλυση διαφορών. Ε, υπάρχουν αρκετές ε, τεχνικές ε, συμφωνίες. Θα πρέπει να δούμε υπάρχει μια πρόταση για τη δημιουργία ενός πάνελ, για μια διαδικασία ενδεχομένως διαμεσολάβησης, mediation θα δούμε, θα πρέπει να συζητηθούν περισσότερο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων τα θέματα αυτά. Ε, ε, ε, έχει γίνει και μία πρόταση να δημιουργηθεί κάτι αντίστοιχο με το Investment Court, αλλά αυτό δεν περιλαμβάνεται όμως στην εντολή. Όσον αφορά γεωγραφική σύνδεξη δεν έχουμε υποβάλει ακόμα κείμενο. Ε, ο Επίτροπος έχει ήδη εκδηλώσει ε, και την πρόθεσή του να ανοίξει και το κεφάλαιο του TST, ε, αλλά ακόμα από τη στιγμή που δεν έχουμε πρόταση δεν μπορούμε να προβλέψουμε και κάποιες κυρώσεις όσον αφορά το ζήτημα του κόστους μεταφοράς και τις εκπομπές στα πλαίσια των ε, συμφωνιών ε, ελεύθερου εμπορίου, FTA, ναι, είναι γεγονός ότι ε, εδώ συμπεριλαμβάνονται, στην Ευρώπη συμπεριλαμβάνονται και το κόστος των εκπομπών και το κόστος των μεταφορών. Για την ώρα δεν έχουμε ακόμα συνολική εικόνα, ωστόσο καλό είναι να δει κανείς ότι οι αυξημένες εκπομπές από την ε, συμφωνία είτε με την Νέα Ζηλανδία είτε με την Αυστραλία ε, μπορούν να μετρηθούν. Είναι μετρήσιμα στοιχεία ε, και η μελέτη αντικτύπου νομίζω ότι βρίσκεται ήδη διαθέσιμη επιγραμμικά. Όταν μιλάμε βέβαια για εκπομπές δεν μιλάμε μονάχα για την, ε, τη μεταφορά αλλά και για τις εκπομπές σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και δυνατότητες χρήσης τεχνολογιών μείωσης των εκπομπών σε καγαστή συνεργασία των δύο πλευρών. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να πω. Όσον αφορά τις, ε, τα safeguards, τα, ε, τις διασφαλίσεις, ναι, απάντηση. Ε, όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, το θέμα των διασφαλίσεων αυτών διασφαλίσεων αυτών ε, θα ληφθεί ε, υπόψη, θα μελετηθεί ακόμα, ε, αποτελεί απλώς μία εναλλακτική ένα ενδεχόμενο. Θα πρέπει να δούμε πώς εντάσσεται το στοιχείο αυτό στο, στο σύνολο, έτσι ώστε το σύνολο να είναι ισορροπημένο και μετά θα αποφασιστούν οι τελικές θέσεις. Ε, ναι, αλλά βέβαια αυτή τη στιγμή ο, ο ελέφαντος στο δωμάτιο ήταν το, το πλοίο. Το πρόβατο. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Μου φαίνεται ότι πρέπει να συνδυάσουμε τις ταχείες αλλά και καλές αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο και δεν πρέπει να περιμένουμε βέβαια μέχρι τελευταία στιγμή Έγκαιρα θα πρέπει να συζητείτε τα κρίσιμα θέματα με τους διαπραγματευτικούς εμπορικούς μας εταίρους και εμείς πρέπει να ενημερωνόμαστε ε, χωρίς να πιέζουμε για την ενημέρωση, ούτω ώστε να υπάρχει απαραίτητη διαφάνεια για να λειτουργεί και η Επιτροπή για να παρακολουθεί. Ναι, πολύ σύντομα. Δεν νομίζω ότι απαντήσατε για την αρχή της προφύλαξης και την ε, αλληλεπίδραση των διαφόρων φορέων ε, συνεργασίας. Η αρχή της προφύλαξης αποτελεί πρακτική, έχει συμπεριληφθεί στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις ως βασική έννοια και υπάρχει στα κείμενά μας και τις προτάσεις μας η μορφή βέβαια που θα λάβει αυτό στην πράξη θα εξαρθεί από τις διαπραγματεύσεις. Και οι διάφοροι ε, φορείς ρυθμιστικής συνεργασίας και πώς αλληλεπιδρούν. Εμείς το εξετάζουμε εδώ και καιρό αυτό το θέμα. Συνήθως είναι προαιρετική βάση. Αυτό μπορούμε να το ενθαρρύνουμε, αλλά όλα εξαρτώνται από την προθυμία των ρυθμιστικών φορέων που καμιά φορά δεν είναι δεδομένη. Και αυτό δεν είναι, είναι θέμα απόφαση τη Κομισιόν. Όχι, αλληλεπίδραση των ρυθμιστικών φορέων συνεργασίας όχι μόνο σε διμερές επίπεδο, δηλαδή αυτό που λειτουργεί μεταξύ δύο χωρών, αλλά ε, ε, ε, αλληλεπίδραση διαφόρων φορέων. Γιατί κάθε σέσε έχει ένα φορέα και υπάρχουν διάφοροι, διάφορες, διάφοροι φορείς που αλληλεπιδρούν. Λοιπόν, καλά, θα το ξαναδούμε το θέμα, λέει ο πρόεδρος. Δεν είναι η τελευταία φορά που τα συζητάμε όλα αυτά. Η κυρία ε, το γνωρίζει αυτό. Ευχαριστούμε τον πρέσβη, την κυρία Κόνιχ και έτσι τελειώσαμε το σημείο 15 και πάμε κατευθείαν στο σημείο 16 που είναι μια πολύ μεγάλη εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία. Κοινή συζήτηση για την Συμφωνία εταιρική Σχέσης ε, Μιλάμε για τα σημεία 16 και 17 στην ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, ε, η διαδικασία διαπραγματεύσεων άρχισε το 2012. Είναι μακρά διαδικασία. Έγιναν και εδώ πολλές συζητήσεις στην Επιτροπή μας. Ε, πήγαν δύο αντιπροσωπείες στην Ιαπωνία, ε, κάναμε ακροάσεις, workshop και είχαμε πάνω από 30 συναντήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης με τη συμμετοχή και πολλών ε, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ε, συνδικάτων κλπ. Έγινε λοιπόν δημόσια συζήτηση πολύ εντατική για την εμπορική αυτή συμφωνία και τώρα είναι έτοιμο το κείμενο. Έγινε στις 9 Ιουλίου μια κρόαση με μεγάλους ε, εμπλεκόμενους και τώρα αρχίζει η διαδικασία κύρωσης. Πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τη συμφωνία. Και ο πρόεδρος και βασικός διαπραγματευτής είναι ο κύριος Πέντρο Σίλβα Περέιρα που λαμβάνει αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα συνάδελφοι. Ελπίζω να περάσατε καλές διακοπές. Σήμερα έχουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων μετά την ε, υπογραφή της ε, συμφωνίας ε, της οικονομικής εταιρικής που έλαβε χώρα τον Ιούλιο, 17 Ιουλίου δηλαδή. Προηγουμένως είχαμε δημόσια ακρόαση εδώ στην Επιτροπή μας, στην ΙΝΤΑ, στις 9 Ιουλίου με τον επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, τεμάτι και διάφορους σημαντικούς παράγοντες τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από την Ιαπωνία. Θα ήθελα λοιπόν εδώ πρώτα απ' όλα να σας πω ότι έχει δημοσιοποιηθεί το κείμενο της συμφωνίας εδώ και λίγους μήνες, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να καθυστερούμε τη συζήτησή μας για την τελική πρόταση και να καταλήξουμε και σε απόφαση. Νομίζω ότι αυτή η σημαντική συμφωνία αξίζει μια πραγματική συζήτηση. Γι' αυτό εξάλλου είχαμε και δύο συναντήσεις της ομάδας παρακολούθησης ήδη τον Απρίλιο και τον Μάιο. Και γι' αυτό και οργανώσαμε και την δημόσια κρόαση όπως σας είπα πριν. μετά την ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε ως εισηγητή σα θα παρουσιάσω πολύ γρήγορα ένα σχέδιο σύστασης που θα συνοδεύεται και από ένα σχέδιο ψηφίσματος. Θέλω εδώ να υπογραμμίσω ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα πρέπει να πάρει μια σημαντική απόφαση τους επόμενους μήνες. Ξέρετε ότι αυτή η συμφωνία είναι μια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα αρχίσει να ισχύει μόνο εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την εγκρίνει. Όμως είναι επίσης σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν εκπλήσει καθόλου το Κοινοβούλιο μας. Εμείς ξεκινήσαμε έγκαιρα νωρίς. Είχαμε ψήφισμα ήδη από τον Οκτώβριο και το 2012 και τα τελευταία χρόνια διάφορες ε, ομάδες παρακολούθησης συναντήθηκαν, 21 μάλιστα. Οπότε το κοινοβούλιο αυτό πάντα στήριζε τις διαπραγματεύσεις. Έχουμε παρακολουθήσει όντως όλη την διαδικασία εκ μέρους των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα πια εμείς πρέπει να αξιολογήσουμε και το αποτέλεσμα στο οποίο κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις. Να ενημερωθούμε από τους διάφορους φορείς και να καταλήξουμε στην τελική μας απόφαση. Η τελική ψηφοφορία θα γίνει στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε να συζητούμε το περιεχόμενο της συμφωνίας αυτής βάσει των δικών της συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Τώρα, ποια είναι κάποια στοιχεία κλειδί που πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας για να αξιολογήσουμε την εταιρική αυτή σχέση. Η στρατηγική διάσταση της συμφωνίας αυτής, η οικονομική ισορροπία των όσων αποφασίστηκαν και ό,τι έχει να κάνει με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρώτα απ' όλα, η στρατηγική σημασία που έχει συμφωνεί αυτή λαμβάνει υπόψη ε, σε ευρύτερα γεωστρατηγικά πλαίσια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία είναι στρατηγικοί εταίροι, συμμερίζονται τις ίδιες αξίες, δημοκρατία, κράτος δικαίου, αλλά και δέσμευση υπέρ της πολυμερούς διάστασης των συστημάτων που διέπουν τη ζωή μας. Από αυτή την άποψη λοιπόν έχει νόημα όχι μόνο να έχουμε μια στρατηγική ε, συμφωνία εταιρική σχέσης, αλλά να ενισχύσουμε και τις διμερείς μας σχέσεις, έτσι ώστε οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας να ανέβουν ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Αυτό βοηθάει την τάξη, το κράτος δικαίου και η συμφωνία αυτή μπορεί να στείλει και ένα σημαντικό μήνυμα για το πόσο μεγάλη σημασία έχει ένα εμπόριο που βασίζεται σε κανόνες, προωθώντας συγχρόνως τις δικές μας προδιαγραφές και αξίες και στην περιοχή της άλλης χώρας, αλλά και γενικότερα. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι η συμφωνία αυτή εταιρική σχέσης είναι πιο σημαντική που, έχει ποτέ, που είχε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πρόκειται για ένα τεράστιο νόγκο και οικονομικά τεράστια σημασία. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι από στρατηγική άποψη είναι πολύ σημαντική αυτή η συμφωνία. Το δεύτερο θέμα τώρα είναι η οικονομική ισορροπία της συμφωνίας αυτής. Η συμφωνία αυτή, χωρίς άλλο, είναι μια φιλόδοξη και συνολική συμφωνία που φροντίζει για να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στις αγορές και να ακολουθούνται κοινοί εμπορικοί κανόνες. Από την έκθεση δικτύπου του 2016 ξέρουμε ότι έχουμε πολλά θετικά στο ΑΕΠ μας από αυτήν την συμφωνία και στο εμπόριο και τα ωφέλη αυτά είναι τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και την Ιαπωνία. Πιο συγκεκριμένα, 97% των δασμών καταργούνται όσον αφορά τις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ιαπωνία. Και διατηρούμε δασμούς για τα πιο ευαίσθητα προϊόντα μας. Η συμφωνία επίσης προστατεύει 205 γεωγραφικές ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι πολύ σημαντικό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μας για την ε, διατροφική βιομηχανία, για την υφαντουργία, ε, τον αμπελοϊνικό τομέα και τα τρόφιμα. Και εδώ θα υποφεληθούμε από μεγάλη μείωση των δασμών. Τώρα, για τους μη δασμολογικούς φραγμούς. Πολλά μη δασμολογικά μέτρα έχουν αντιμετωπιστεί από την Ιαπωνία και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, αλλά σίγουρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην παρακολούθηση η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να καταργήσει το 10% των ε, δικών της ε, δασμών ε, στοχήματα και αλλού για 10 χρόνια ενώ η Ιαπωνία δεσμεύτηκε να ακολουθήσει ακόμα περισσότερο τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Οπότε πρόκειται για μια συμφωνία από την οποία έχουν να κερδίσουν και οι δύο πλευρές. Η Ιαπωνία επίσης όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Θα φροντίσει να καταργήσει την ε, δικλίδα ασφάλειας. Οπότε θα καταλήξουμε να έχουμε μία κατάσταση στην οποία θα υπάρχει απολύτως ίση μεταχείριση. Τώρα η αυτή αυτή συμφωνία με την Ιαπωνία φυσικά περιλαμβάνει και το εμπορικό κεφάλαιο, όπου επιβεβαιώνουν οι δύο πλευρές τη δέσμευσή τους για διμερείς συμφωνίες και όσον αφορά το κλίμα και το περιβάλλον αλλά και την ε, βιωσιμότητα. Η συμφωνία περιλαμβάνει και καινοτόμα συστατικά, ένα κεφάλαιο για τη διακυβέρνηση, ένα κεφάλαιο που αναφέρεται στη δέσμευση υπέρ ε, της Συμφωνίας των Παρισίων και επίσης όπως συμβαίνει και με τον Καναδά εδώ υπάρχει δέσμευση για να ακολουθούμε τις προδιαγραφές του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Αυτό το καλωσορίζουμε βέβαια. Όμως γνωρίζουμε ότι η Σύμβαση 105 και 111 που έχει να κάνει με τις διακρίσεις όσον αφορά την απασχόληση και το δικαίωμα εργασίας δεν έχουν κυρωθεί ακόμα από την Ιαπωνία. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως ο σεβασμός των συμβάσεων αυτών είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε να επιμένουμε ελπίζοντας να υπάρξει πρόοδος από πλευρά της Ιαπωνίας και να κυρώσει αυτές τις δύο συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Ξέρω, πρέπει να ολοκληρώσω, Πρόεδρε, οπότε να προσθέσω μόνο ότι το κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη θα μας επιτρέψει να καταπολεμήσουμε την παράνομη ελεία και την παράνομη υλοτομία. Ξέρουμε ότι είναι πολύ ισχυροί μηχανισμοί της Ιαπωνίας. Πάντως μετά από το έτοιμά μας, η συμφωνία περιλαμβάνει και ρήτρα αναθεώρησης για το κεφάλαιο βιωσιμότητας, που επιτρέπει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο αυτό το κεφάλαιο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προσβεί σε αυτήν τη ρήτρα σε εφόσον χρειαστεί. Ολοκληρώνοντα, Πρόεδρε, όλοι γνωρίζουμε ότι η συμφωνία αυτή δεν περιλαμβάνει κάτι για την προστασία των επενδύσεων. Θα γίνουν χωριστές διαπραγματεύσεις γι' αυτό και για την ροή δεδομένων Υπάρχει και εδώ μια ρήτρα αναθεώρησης. Τρία χρόνια μετά. Οπότε θα πρέπει να έχουμε διευκρίνηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με αυτές τις δεσμεύσεις. Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας και προσβλέπω στα σχόλιά σας για να ετοιμάσουμε την πολιτική μας απόφαση. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστούμε πολύ εισηγητές. Τώρα δύο λεπτά ο καθένας. Ο κύριος Κολέτη είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ κύριος Βαλές. Θα βελτιωθεί το εμπόριο στα αγαθά και τις υπηρεσίες και θα βελτιωθούν και οι επενδύσεις. Εκατέρωθεν κάποια στοιχεία. 99% των δασμών που πληρώνουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες που εξάγουν στην Ιαπωνία θα καταργηθούν 85% της παραγωγής στην Ευρώπη θα εισάγεται χωρίς δασμού στην Ιαπωνία. Η συμφωνία αναγνωρίζει το ειδικό καθεστώς και προστατεύει ε, στην Ιαπωνική αγορά πάνω από 200 γεωργικά προϊόντα από διάφορες γεωγραφικές προελεύσεις. Οι εταιρείες οι ευρωπαϊκές θα μπορούν ισότιμα να συμμετέχουν στη, στους διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις σε 48 βασικές πόλεις στην Ιαπωνία. Ε, δεν υπάρχουν εμπόδια επίσης στις συμβάσεις στους σιδηροδρόμους. Η Συμφωνία Στρατηγικής Συμφωνίας θα βελτιώσει τη συνεργασία ε, και σε άλλους τομείς πέρα από το εμπόριο όπως ασφάλεια και άμυνα, ενέργεια και κλίμα και ανταλλαγές ανθρώπων. Ε, επίσης η συμφωνία είναι σαφές πολιτικό μήνυμα ε, υπέρ των ελεύθερων συναλλαγών και κατά του προστατευτισμού βλέποντας κυρίως τι γίνεται στη ΗΠΑ. Τονίζω με έμφαση τη σημασία και στρατηγική σημασία δεδομένων των διεθνών συνθήκων ε, αυτής της συμφωνίας. Επίσης, ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, και την πολιτική της Κίνας, μια ζώνη ένας δρόμος. Ε, με την Ιαπωνία έχουμε κοινέ αξίες πολλές και αυτή η συμφωνία αναμενόταν για πολύ καιρό. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να συνενέσουμε σύμφωνα και το ταχύτερο δυνατόν να δώσουμε την έγκρισή μας για τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Η ΕΜΑ. Εξ ονόματος των Σκιώδους Ισιάρα ε, που δεν μπόρεσε να ήθελε να δεν μπορούσε να έρθει Πρέπει να πω ότι αυτή είναι συμφωνία ορόσημο. Η εφαρμογή της συμφωνίας εταιρική σχέσης θα αυξήσει τις δυνατότητες εξαγωγών για τις επιχειρήσεις μας, θα βελτιώσει τον ανταγωνισμό, θα δημιουργήσει οικονομική ανάπτυξη, θα βελτιώσει τους καταναλωτές μειώνοντας τις τιμές και των βασικών αγαθών και των υπηρεσιών. Είναι στρατηγική σημασία. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία δείχνουν ότι είναι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου. Τώρα που είναι τόσο διαφορετικά τα πράγματα από ε, άλλους, ε, εμπλεκο, άλλους παίκτες στην αγορά. Ε, υπάρχει ε, η, δυνατό, το, η δυνατότητα ανοίγματο των αγορών στην Ιαπωνία σε παραδοσιακούς τομείς όπως κρέας, γαλακτοκομικά, ε, παπούτσια και ε, ένδυση που παλιά ήταν προστατευμένα. Ε, τώρα μπαίνουμε και στις δημόσιες αγορές και στους σιδηροδρόμους στην Ιαπωνία ε, με την ε, ρήτρα επιχειρησιακής ασφάλειας. Μπορούμε έτσι να παραδίδουμε ε, σε έναν αριθμό πόλεων προϊόντα. 110 θα είναι οι γεωγραφικές ενδείξεις στα προϊόντα και πιστεύουμε ότι η βιομηχανία μας θα ωφεληθεί Ε, η συμφωνία θα ωφελήσει την Ευρώπη. Ε, ε, επίσης, η συμφωνία θα οδηγήσει στην κατάργηση πολλών ρυθμιστικών φραγμών πρόσβαση στην Ιαπωνική αγορά. Ε, τη χαιρετίζομαι. Σε κάποιους τομείς μπορούσαμε να είχαμε προχωρήσει περισσότερο. Ε, για παράδειγμα, το ECR θα ήθελε φιλόδοξες ε, προτάσεις και διατάξεις για την ροή των δεδομένων. πάντως, στηρίζομαι τις παράλληλες διαπραγματεύσεις ε, διότι έτσι θα διευκολυνθεί η ψηφιακή οικονομία. Το ECR συμφωνεί με την απόφαση του ε, Συμβουλίου. Ελπίζουμε να οριστικοποιηθεί η συμφωνία σύντομα και θα συνεργαστούμε και με τον εισηγητή και με τους σκιώδεις. Ο Κλάους Μπούχνερ για τους πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ. Για τις υπηρεσίες, αυτό το κοινοβούλιο ήδη εξέφρασε ανησυχίες πολλές φορές σχετικά με τους αρνητικούς καταλόγους. Ακόμα πιο σημαντικό, η τελική έκθεση της Επιτροπής Πάναμ σε αυτού του κοινοβουλίου συνέστησε ε, τα κεφάλαια επενδύσεων των, συμφωνι... των ΣΕΣ να διαπραγματεύονται με βάση θετικούς καταλόγους. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια αντίφαση σε σχέση με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεύτερο πρόβλημα, το κεφάλαιο για το εμπόριο και την βιώσιμη ανάπτυξη. Η Ιαπωνία δεν έχει κυρώσει δύο βασικές συμβάσεις ε, του ΔΟΕ. Ελπίζω και το ε, ε, Γκούε να τα πει αυτά, γιατί εγώ δεν έχω πολύ χρόνο. Τονίζω όμως και το θέμα της ξυλίας. Ε, στο, στην ακρόαση του Ιουλίου μάθαμε ότι υπάρχει νομοθεσία για την, ε, τις προϋποθέσεις δέουσας ε, επιμέλειας στην Ιαπωνία. Ε, αυτή, αυτή η νομοθεσία έχει εξεταστεί, μοιάζει με τη δική μας πότε θα τεθεί πλήρως σε ισχύ αυτή η καινούργια νομοθεσία. Η αρχή της προφύλαξης εδώ συνιστά μεγάλο πρόβλημα. Η Ιαπωνία έχει κάποια νομοθεσία σε αυτό το τομέα, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν επαρκεί. Ήθελα να σας θυμίσω την καταστροφή στην Ιαπωνία στο Κόντεγκάν που οφειλόταν ακριβώς στην ε, μία εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης. Για τη ροή των δεδομένων εμείς έχουμε μία απόφαση ε, με την Ιαπωνία ήδη. Γιατί να ξανανοίξουν οι διαπραγματεύσεις ε, σχετικά με τις διατάξεις ροής δεδομένων στην ΣΕΣ. Τέλος, η Κομισιόν έχει ανησυχίες σε σχέση με την ε, πολιτική ε, των συντελεστών γιατί η Ιαπωνία σε ορισμένα βασικά θέματα είναι B-. Να σας... Ε, δεν είναι η ΣΕΦΤΑ, είναι η TIPA. Είναι η η Οικονομική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης με την Ιαπωνία. και ο κύριος Σόλτς για την ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τη διόρθωση. Είπατε ότι πρόκειται για συμφωνία εταιρικής, ε, εταιρική σχέση. Ε, είναι πολιτική όμως η συμφωνία που περιλαμβάνει πολύ σημαντικά οικονομικά θέματα. Ε, οι περισσότερες ομάδες εκφράστηκαν θετικά εγώ θέλω λίγο να ε, δω πιο κριτικά το ζήτημα γιατί υπάρχουν πολλές διμερείς εμπορικές συμφωνίες ε, πρόσφατα ε, συνήφθησαν και πάντοτε συζητούσαμε για το θέμα το ρυθμιστικό. Είναι σημαντικό, είναι και είναι σωστό, ότι στο κομμάτι ΕΖΕΣ, δηλαδή ελευθέρων συναλλαγών ε, δεν έχουμε πολλές αρμοδιότητες για τις κοινέ επιτροπές. Υπάρχει μια μεγάλη γκρίζα ζώνη σχετικά με τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες ε, και τη σχέση ε, των Επιτροπών με τους δημοκρατικούς θεσμούς που είναι υπεύθυνοι για την ρύθμιση αλλά και για το νομοθετικό πλαίσιο. Γι' αυτό ε, το ζήτημα αυτό δεν έχει επιληθεί επαρκώς. Οι εξελίξεις θα δείξουν σε ποιο βαθμό θα υπάρξει πρόβλημα. Δηλαδή οι εμπορικές ροές, οι σχέσεις οικονομικής συνεργασίας, ε, αν θα ε, ωφεληθούν ε, από το σύστημα αυτό ή αν ο ανταγωνισμός και συζητήσαμε για την πολιτική ανταγωνισμού προηγουμένως ε, θα είναι η μοναδική παράμετρος που θα λαμβάνεται υπόψη πράγμα που δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας αλλά και ελλειπούς εμπιστοσύνης από την πλευρά του κόσμου. Κάτι άλλο που πάει προς την ίδια κατεύθυνση είναι οι ε, δημόσιες συμβάσεις και Ε, οι δύο πλευρές ε, έχουν την ε, αρχή του γενικού ενδιαφέροντος, επίσης ότι δεν θα υπάρξει ιδιωτικοποίηση, αλλά υπάρχει σαφώς η δυνατότητα να υπάρξει μια γκρίζα ζώνη ε, και όταν υπάρξει ένα διαγωνισμός να ε, δημιουργηθεί αβεβαιότητα. Δεν μπορεί να υπάρχουν προβλήματα δηλαδή. Επίσης, ε, το 7-2 αυτό είναι ανοιχτό σε σχέση με την προστασία που παρέχεται και σε σχέση και με τη Συμφωνία του Ειρηνικού. Ε, υπάρχουν εκεί ορισμένα ζητήματα που αφορούν τη διαιτησία ε, και επίσης ε, το αν θα μπορούν να παρεμβαίνουν τα δικαστήρια των χωρών. Αυτό είναι ακόμα κάτι που πρέπει να ρυθμίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ρενά, ευχαριστώ πολύ. Ίσως υπάρχει και μία διαφωνούσα φωνή σε σχέση με τα όσα είπε και ο εισηγητής προηγουμένως. Πρώτον, ερωτήσεις μάλλον προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το κεφάλαιο ε, για την βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, στα πλαίσια του ε, TPP είχε η Ιαπωνία υπογράψει ένα σχετικό κεφάλαιο. Γιατί λοιπόν δεν επέμεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να υπάρχει ένα κεφάλαιο κατά αυτή την έννοια αλλά με κυρώσεις. Ξέρω ότι η Κομισιόν δεν ήθελε κάτι τέτοιο, ε, επίσης δεν ήθελε ένα κεφάλαιο για το SDS ε, και ε, αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Δεύτερη ερώτηση για το χρηματοδοτικό των χρηματοπιστωτικών θεμάτων. Είναι πιο επιφυλακτική η Ιαπωνία όσον αφορά την απελευθέρωση και διάβασα προσεκτικά ότι η Ιαπωνία έχει επιβάλει κάποιες, έχει αναφέρει κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά ε, τι, τα χρηματοπιστωτικά ενώ ε, ε, η Κομισιόν όχι. Ζητώ λοιπόν από την Κομισιόν να είναι πιο προσεκτική λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα συνέβησαν πριν την κρίση του 2008. Επίσης εγώ πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα παρά να γίνει παραπομπή σε κάποιες συμβάσεις να, να είχε ζητηθεί η επικύρωσή τους πριν από την υπογραφή της συμφωνίας. Επίσης θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη ε, προσοχή όσον αφορά την ε, δέουσα επιμέλεια, due diligence, γιατί ξέρουμε ότι στην Ασία και στην Ανατολική Ασία ε, η Ιαπωνία είναι από, τις πιο, από τους πιο κακούς μαθητές όσον αφορά την αποψήλωση των δασών. Έπρεπε να είμαστε πιο προσεκτικοί λοιπόν. Ακούμε επίσης ότι έχουμε επιτέλους μια συμφωνία που η ε, που είναι η καλύτερη συμφωνία όσον αφορά ε, τη, ε, τη Συμφωνία των Παρισίων. Αλλά ο οργανισμός για, του Νικολάου Λό αναφέρει ότι πρόκειται για κλιματοκτόνο συμφωνία. Πρόκειται για κλιματοκτόνο και όσον αφορά την αποψήλωση που ανέφερα προηγουμένω των δασών και όσον αφορά την αναρχία αλληλεία κλπ. Νομίζω ότι αν δεν είχε ήδη παρετηθεί ο Νικολάου Λό θα το τώρα βλέποντας τη συμφωνία αυτή. Ίσως, ε, ίσως ε, βάσει της συμφωνίας αυτής ε, να δημιουργηθεί ε, ανάπτυξη 0,04% αλλά με ποιο τρόπο θα ήθελα να μάθω εγώ παρόλα αυτά λαμβάνουμε υπόψη την αποψήλωση των δασών, τον υπολογισμό του κόστους των μεταφορών κλπ. Αυτή η ρήτρα αναθεώρησης δεν θα λύσει τα πάντα. Στην ΣΕΤΑ ας πούμε υπάρχει τέτοια ρήτρα όπου αναφέρεται όμως ότι δεν θα δοθεί ε, το πράσινο φως ε, στο, στη δική μας πλευρά σε περίπτωση ε, που τα θέματα φτάσουν ενώπιον των δικαστηρίων. Ευχαριστώ πολύ Καρολίνα. Ευχαριστώ. Ε, θέλω να πω ότι το ΣΕΤΑ είναι μια α, συμφωνία που ε, χρησιμεύσε ε, ως ε, πρότυπο για τις μελέτες μας. Επίσης επελέγει μια αρνητική προσέγγιση και το θέμα της προστασίας είναι διαφορετικό από ό,τι στη ΣΕΤΑ. Βεβαίως υπάρχουν πολλές ερμηνευτικές επεξηγήσεις στη ΣΕΤΑ. Δεν υπάρχει αυτό στην συμφωνία αυτή της ΣΕΣ. Ε, επίσης για το, τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος έχουν αποδυναμωθεί πιστεύω γιατί ε, αν δούμε τη συμφωνία ε, στα πλαίσια του ΠΟΕ δεν υπάρχει συνέχεια, υπάρχει μια αντίφαση. Έχει αποδυναμωθεί το κείμενο σε σχέση με τις άλλες, το κείμενο άλλων συμφωνιών. Το Κοινοβούλιο ε, θα πρέπει ε, να δραστηριοποιηθεί οι εκπρόσωποι πώς διορίζονται και πώς μπορεί να παρακολουθεί το έργο του στο Κοινοβούλιο. Ε, και αυτό είναι σημαντικό για το ρόλο μας. Είναι σημαντικό να υπάρχουν και δυνατότητες ή η Ιαπωνία να συμφωνήσει με μια καλύτερη ε, συμφωνία που θα περιλαμβάνει και θα ενσωματώνει περισσότερες δικές μας προτάσεις. Ευχαριστώ. Ιαν Μαρή Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτό το καλοκαίρι προχώρησε η συμφωνία με την Ιαπωνία ε, χωρίς ε, προηγουμένως να δώσει την έγκρισή του στο την του κοινοβουλευτικό σώμα και μετά το Συμβούλιο, η συζήτηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να φροντίζει να προστατεύει τους θεσμούς. Πολύ ωραία, αλλά αυτά τα οποία ε, προτείνονται εδώ πέρα δεν υπάρχουν στη συμφωνία με τη Σιγκαπούρη. Για τα δεδομένα, για παράδειγμα. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνεται. Υπάρχει αγωνία ότι δεν θα καλύψει αυτό το οποίο θέλουμε αυτή η συμφωνία. Μία συμφωνία η οποία σπρώχνει τελικά τους ε, Ευρωπαίους πολίτες να δεχτούν πράγματα και είναι ουσιαστικά σαν να πυροβολούμαστε στα πόδια εμείς η Επιτροπή μας. Πάντω δεν πρόκειται μόνο για τα προσωπικά δεδομένα, πρόκειται και για τη διατησία. Οπότε αυτό που εγώ έχω να συμβουλεύσω τόσο τον εισηγητή όσο και την Επιτροπή είναι να φροντίσουν πρώτα να τηρηθεί η διαδικασία για τη λήψη αποφάσεων και να ενημερωθεί ο κόσμος πριν περάσει και από το κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Και τώρα Θα δώσω το λόγο στον κύριο και ο οποίος ε, είναι ε, ο επικεφαλής ε, τη της του Κοινοβουλίου για τη σχέση με την Ιαπωνία. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω δύο σχόλια, ένα εξειδικευμένο και ένα γενικό. Πρώτον, για να αντιδράσω σε όσα αναφέρθηκαν για τις συστάσεις της Επιτροπής για τα Panama Papers σχετικά με, με την αρχή της, του θετικού καταλόγου Positive List Principle. Ε, μπορώ να υπενθυμίσω ότι αυτό ε, σχετίζεται με κεφάλαια χρηματοπιστωτικά και στόχος του αιτήματο αυτού ήταν μονάχα η πραγματική οικονομία να έχει ε, την απελευθέρωση που χρειάζεται και να μην αναφερθούμε λοιπόν στην ε, φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή, αλλά η Ιαπωνία δεν φημίζεται ως φορολογικός παράδεισος, άρα δεν υπήρχε λόγος. Ο Πέτρος Σίλβα Περέιρα πολύ καλά τα είπε γενικά, πάντως είναι σαφές και από όλε τις μελέτες και, ε, και αν δει κανεί τα πράγματα και από πλευράς επιχειρήσεων και από πλευράς των πολιτών, οπωσδήποτε ε, η συμφωνία αυτή θα είναι για όλους επωφελής και οπωσδήποτε ε, θα αποτελέσει και συγκολητική ουσία έτσι ώστε να προωθηθούν ακόμα περισσότερο οι σχέσεις μας. Στο σημερινό κόσμο, στον κόσμο στον οποίο ζούμε, νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, ε, εξετάζοντας την συμφωνία από όλες τις πλευρές, μόνο θετικά μπορώ να βρω. Ίσως ε, κάποιοι συμμετέχοντες ε, της, ε, στην εσωτερική αγορά θα έχουν ίσως μεγαλύτερο πρόβλημα προσαρμογής στους νέους κανόνες. Και το λέω ξέροντας, ε, έχοντας περάσει την ε, μισή ζωή μου σε ε, οικονομία που δεν είναι οικονομία αγοράς, παρ' όλα αυτά διαπιστώνω ότι μόνο με το σωστό ανταγωνισμό μπορεί να προχωρήσει η οικονομία. Υπάρχουν στοιχεία της συμφωνίας που είναι πολύ σημαντικά και ευελπιστώ ότι θα γίνει μια διαφανής συζήτηση, δηλαδή συζήτηση με όρους διαφάνειας ε, και θα ολοκληρωθεί θετικά ε, και οπωσδήποτε σε τούτη τη θητεία το θέμα αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ από την Κομισιόν ο κύριος Μάρκο Τσιρούλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους. Και ευχαριστώ όλους τους βουλευτές, μέλη τούτης της Επιτροπής για τα ενδιαφέροντα σχόλια τα οποία ε, εξέφρασαν και τα οποία εμείς ε, σημειώνουμε προσεκτικά. Θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένες από τις ερωτήσεις ε, που και τα σχόλια, ορισμένα από τα σχόλια που ακούστηκαν. Υπάρχει ένα συχνό ερώτημα. Είχα μάλιστα παρόμοια συζήτηση και στην Επιτροπή ΕΜΒΗ σχετικά με την αρχή της πρόληψης και νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα όταν μιλάμε ε, για ρήτρα ε, πρόληψης. Ναι, είναι γεγονό ότι στο κεφάλαιο TST ε, αναφέρεται κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτή ε, η αρχή ε, συμπεριλαμβάνεται στις συμφωνίες μας. ως γενική αρχή που μπορεί να προσαρμοστεί σε πολλές περιπτώσεις μεταξύ των οποίων και τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα πάντα ευθυγραμμίζονται ε, απολύτως ας πούμε με τις υφιστάμενες ε, διατάξεις του, ε, για την ασφάλεια των τροφίμων καθώς επίσης και με τις δευτερογενείς διατάξεις και δευτερογενή κείμενα για τις ορμόνες ή για για, τις, ε, για τα μεταλλαγμένα. Οπωσδήποτε λοιπόν μπορώ να πω ότι τίποτα δεν ε, μας προβληματίζει ας πούμε όσον αφορά την, χρήση, την αναφορά της αρχής της πρόληψης και ότι οπωσδήποτε παρέχονται και όλα τα απαραίτητα εχέγγυα τα οποία θα ε, τα οποία ε, πηγαίνουν ας πούμε με, μαζί με την αρχή της πρόληψης ε, ας πούμε στο κεφάλαιο SPS και στο κεφάλαιο για το περιβάλλον καθώς επίσης και στο ειδικό άρθρο για τις εξαιρέσεις που εφαρμόζεται πλήρως όλα αυτά αναφέρονται ιδιαίτερα προσεκτικά. Πρόκειται για μια αρχή η οποία προστατεύεται στη συμφωνία όσον αφορά την υλοτομία. η, ε, η Ιαπωνική νομοθεσία στη δημιουργία της οποίας έχει συμβάλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα εγκρίθηκε αλλά ήδη εφαρμόζεται ε, και ε, εργαζόμαστε στενά με την Ιαπωνική πλευρά έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης εφαρμογή καθώς επίσης και ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας. Ε, και πρέπει να σας πω ότι όχι μονάχα ε, εφαρμόζεται ήδη η νομοθεσία αλλά εφαρμόζεται και η αρχή της εδέουσας επιμέλειας έτσι ώστε ε, να, να μην υπάρχει περίπτωση εισαγωγής παράνομα υλοτομημένου υλικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και ε, εν πάση περιπτώσει όσον αφορά αυτά τα θέματα παραμένει αμετακίνητη η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ε, νομοθεσία της. Ε, ναι, όσον αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη και την παρατήρηση που ακούστηκε, ναι βεβαίως το σημειώνουμε και είναι ένα θέμα το οποίο επανειλημμένα έχει προκύψει στις συζητήσεις και το συμπεριλαμβάνουμε κατά κανόνα στις εμπορικές μας ε, συναλλαγές. Ε, όπως άλλωστε και για τα θέματα τα οποία σχετίζονται ε, με τον ΔΟΕ και την Καναδά ή την Αυστραλία και εδώ προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας. Προς ώρας σημειώνουμε τα σχόλιά σας όσον αφορά τώρα άλλα θέματα τα οποία γέρθησαν εδώ, ας πούμε για τις υπηρεσίες. Ναι, η διαπραγμάτευση ε, βασίζεται σε αρνητική προσέγγιση ε, για ε, ε, ευαίσθητα θέματα. Ναι, μπορεί κανείς να διαλέξει τη μία, τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μετράει είναι η ουσία. Το θέμα είναι εάν προστατεύουμε εμείς τους ευαίσθητους τομείς μας, εάν προωθούμε άλλους ευαίσθητους τομείς, δηλαδή που παρουσιάζουν άλλη μορφή ευαισθησίας. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να μας απασχολούν και πρέπει να απασχολούν φαντάζομαι και τα μέλη εδώ. Ε, και οπωσδήποτε απασχολούν την κοινή γνώμη και η απάντηση γιατί πρέπει να είμαι σύντομος, ε, είναι αυτή, αλλά βεβαίως μπορώ να σας δώσω και αγραπτά αν θέλετε. Ε, και η σύντομη απάντηση είναι ότι οι υπηρεσίες προς το, για το δημόσιο καλό, για το κοινό καλό, οπωσδήποτε προστατεύονται. Και επίσης και σε ε, αντίστροφη περίπτωση ε, εάν αποφασιστεί δηλαδή η απελευθέρωση ε, μπορεί να αντιστραφεί η διαδικασία με την Ιαπωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Σύντομα αν μπορεί ο εισηγητής μας να εξάγει κάποια συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Μίλησα ήδη αρκετά. Οπότε απλώς θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέρφους για τις παρατηρήσεις τους θα τις λάβω υπόψη μου στο σχέδιο κειμένου που θα ετοιμάσω και θα σας το παρουσιάσω σύντομα. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διευκρινήσεις που έδωσε. Θα έχουμε και αποστολή της ΙΝΤΑ 18 με 20 Σεπτεμβρίου στην Ιαπωνία. Οπότε έτσι έχουμε άλλη μια ευκαιρία να εκφράσουμε τις απόψεις μας απευθείας σε διάλογο με τους Ιάπωνες εταίρους. Κυρίως όσον αφορά την ε, κύρωση από αυτούς των συμβάσεων του ILO, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε στους Ιάπωνες ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ αν προχωρούσαν σε αυτή την κύρωση. Προσβλέπω σε καλή συνεργασία με τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. 27 Σεπτεμβρίου θα ξανασυζητήσουμε για αυτό το θέμα. Ωραία. Και έτσι τελείωσε και αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ήταν τα σημεία 16 και 17 και τώρα πάμε στο σημείο 18. Η συμφωνία με το Μαρόκο, εμπορική συμφωνία με το Μαρόκο που προσπαθούμε να πετύχουμε. Είναι κάτι που έχουμε συστήσει αρκετές φορές. Θα πάει και την προσωπία σύντομα στο Μαρόκο και στη Δυτική Σαχάρα. ξέρουμε τις διαφορετικές απόψεις, την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και μετά από διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο η Επιτροπή παρουσίασε μία νέα πρόταση. Ήρθε και ο Επιτροπός μας, ο κύριος Μοσκοβισή, που θα μας εξηγήσει αυτήν τη νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε να έρθω για να ανταλλάξουμε απόψεις για αυτό το σημαντικό ζήτημα, που είναι και ευαίσθητο. Και σίγουρα χρειάζεται ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Ιουνίου ενέκρινε πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για συμφωνία με το Μαρόκο που τροποποιεί τη συμφωνία σύνδεσης με τη χώρα αυτή προκειμένου να υποφεληθεί από δασμολογικές προτιμήσει η Δυτική Σαχάρα. Το Συμβούλιο στις 16 Ιουλίου ενέκρινε την απόφαση για την υπογραφή της συμφωνίας αυτής και την ίδια μέρα ενέκρινε και την απόφαση ε, σχετικά με τα συμπεράσματα, την κατάληξη της συμφωνίας. Οπότε έγινε εκεί η έγκριση αυτή. Τώρα γίνονται άλλες συζητήσεις τώρα για την αλληλευτική συμφωνία. Ξέρετε ότι είναι του συναδέλφου Βέλα αρμοδιότητα τα αλληλευτικά, οπότε θα τα αφήσω γι' αυτόν. Τώρα, εμείς θα ανταλλάξουμε απόψεις για διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δασμολογικά και μπορώ να σας πω ότι ανταποκρίνονται σε τρεις στόχους, με τους οποίους νομίζω όλοι συμφωνούμε. Πρώτον, η υποχρέωση συμμόρφωσης με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Δεκεμβρίου του 2016. Για μας αυτός ήταν ο χάρτης πορείας μας από την αρχή. Δεύτερον, τη φιλοδοξία μας υπέρ της Δυτικής Σαχάρας για τις δασμολογικές προτιμήσεις. Και νομίζω ότι είναι κάτι με το οποίο συμφωνούμε όλοι και η Επιτροπή. Και το τρίτο, υπήρχε μια υποχρέωση να μην αναμειχθούμε στην πολιτική διαδικασία, γιατί θέλαμε να είμαστε ρεαλιστές. Όταν υπάρχει ένα νομικό ζήτημα, είναι νομικό και δεν θα έπρεπε να υπάρχει πολιτική παρέμβαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν προσπάθησε να αποφύγει κάθε ερμηνεία η οποία θα οδηγούσε σε αλλαγή θέσης ή άποψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τροποποίηση της συμφωνίας δεν έχει σαν στόχο να αποφασίσει ποιο θα είναι το καθεστώς της Δυτικής Σαχάρας τελικά. Όχι, αυτό είναι θέμα του ΟΗΕ, είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Και η συμφωνία αυτή έγινε χωρίς να προκαταλαμβάνονται οι θέσεις του Μαρόκο ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το καθεστώς της Δυτικής Σαχάρας. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό και γι' αυτό ήθελα να το έχω ξεκαθαρίσει ευθύ αρχή. Αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο δεν συζητάμε σήμερα. Είναι το ΙΕ όπω είπαμε. Ο δικός μας στόχος, που ήταν πολύ συγκεκριμένος, ήταν ε, η νομική και η οικονομική διάσταση, έτσι όπως τίθεται από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και αυτό προσπαθήσαμε και εμείς να πετύχουμε. Τα υπόλοιπα είναι για τον ΟΓΕ. Η πρόταση αυτή, λοιπόν, περιλαμβάνει μια τεχνική λύση για να ε, δώσουμε απάντηση στις ανησυχίες του δικαστηρίου από την απόφασή του το 2016 να υπάρχουν δηλαδή οικονομικά ωφέλη για τη Δυτική Σαχάρα από τις συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ περίπλοκο και πολιτικά και νομικά αυτό το ζήτημα και γνωρίζω πολύ καλά τι διακυδεύεται. Και τα ξέρει αυτά και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Συνεργαστήκαμε λοιπόν για να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους. Είμαι πεπισμένος Λοιπόν, και με την κυρία Μογκερίνη, η οποία έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα αυτό, ότι το κείμενο της 16ης Ιουλίου του Συμβουλίου είναι και η καλύτερη δυνατή απάντηση που μπορούμε να δώσουμε. Αυτό είναι σαφές. Υπογραμμίζουμε επίσης ότι δείχνοντα το σεβασμό μας στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρότεινε προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας. Σας αφήνουμε τη δυνατότητα να αποφασίσετε πρώτα, οπότε μετά την απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου του 2016 τα προϊόντα της Δυτικής Σαχάρας δεν χαίρουν δασμολογικής προτίμησης προς το παρόν. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να αναφερθώ σε τρία στοιχεία κλειδί. Πρώτον, συμμόρφωση με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και οργάνωση των διαβουλεύσεων με τον πληθυσμό της Δυτικής Σαχάρας. Μέσα σε ένα πολιτικό πλαίσιο ιδιαίτερα περίπλοκο λοιπόν, το δικαστήριο δεν έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα πετύχουμε τη συνένεση του ντόπιου πληθυσμού. Μπορώ όμως να σας διασφαλίσω και αυτή είναι και η άποψη των νομικών υπηρεσιών τόσο της Επιτροπής όσο και του Συμβουλίου ότι όλα τα μέτρα είναι δυνατά προκειμένου να εφαρμόσουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Προβλέπεται λοιπόν διαβούλευση ευρεία με τη συμμετοχή όλων των ε, κατοίκων της Δυτικής Σαχάρας και με το Πολυσάριο, τους οικονομικούς φορείς, που ως επιτοπλίστων τάχθηκαν υπέρ της συμφωνίας. Θελήσαμε να έχουμε μια ουδέτερη προσέγγιση, χωρίς πολιτική διάσταση. Φροντίζοντας να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη συμμετοχή. Επευθεθήκαμε σε όλες τις οργανώσεις, σε όλους τους εκπροσώπους, ώστε να έχουμε όσο γίνεται ευρύτερη βάση συμμετοχής. Τώρα κάποιοι δεν θέλησαν να συμμετάσχουν. Το σέβομαι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό. Αλλά το λέω γιατί θα τεθεί ότι εμείς τίναμε χείρα και έγιναν όλες οι προσπάθειες ώστε να έρθουν όλες οι οργανώσεις στις ε, συναντήσεις που είχαμε. Συνεχίζουμε να ακούμε το κόσμο, να ακούμε προτάσεις, οπότε είμαστε στη διάθεση όλων. Και το Πολυσάριο. Ζητήθηκε η γνώμη του. Είμαι πεπισμένος ότι πρόκειται για μια πολιτική απάντηση και νομικά εύστοχη που προτείνει το δικαστήριο για τον πληθυσμό της Δυτικής Σαχάρας. Δεύτερον, ποιες θα είναι οι εξελίξεις στη Δυτική Σαχάρα. Σήμερα τα προϊόντα από εκεί δεν εποφελούνται, όπως είπαμε, από δοσμολογικές προτιμήσεις, άρα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με άλλα προϊόντα που μπορούν να επωφεληθούν από αυτές. Δεν υπάρχει λοιπόν ίση αντιμετώπιση, κάτι το οποίο αντιβαίνει με τις αρχές μας. Επιπλέον, η έκθεση για τα ωφέλη του τοπικού πληθυσμού που ετοίμασαν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λένε ότι πρέπει το ωφέλη να πηγαίνουν εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Τώρα πιο συγκεκριμένα, περιμένουμε ένα θετικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες επιτόπου στη Γεωργία, στην Αλία. Έχουμε 14.000 ανθρώπους που εξαρτώνται από τη Γεωργία και έχουμε 65 εκατομμύρια ευρώ από προϊόντα που εξάγονται στη Γεωργία και 100 εκατομμύρια από την Αλία. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μεγάλα ποσά δασμοί που κερδίζονται με τις δρομολογικές προτιμήσεις είναι λίγο παραπάνω από 6 εκατομμύρια για τα γεωργικά προϊόντα και 9 παραπάνω από 9 για την αλία. 15 εκατομμύρια δηλαδή συνολικά. Καταλαβαίνετε ότι τα ποσά αυτά στην τοπική οικονομία έχουν τεράστιο αντίκτυπο. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι να νηθούμε στα πρώτα Δυτική Σαχάρας ε, τις δασμολογικές προτιμήσεις είναι κάτι το οποίο πλήττει τα προϊόντα της περιοχής και κυρίως τα λιευτικά, που όπως είδαμε είναι αποφασιστική σημασία για την οικονομία της περιοχής. Έτσι καταλαβαίνετε ότι οι συνέπειες είναι αρνητικές επί του πληθυσμού και δημιουργούν ε, κάποια επιπλέον αδυναμία στην περιοχή. Αν δοθούν τέτοιες ε, δασμολογικές προτιμήσεις, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και επενδύσεις, απασχόληση. Η έκθεση πολύ συγκεκριμένα αναφέρει τους στόχους. Οι πηγές μας είναι όχι μόνο από το Μαρόκο, Εννοείται ότι και εκεί παρακολουθήσαμε την κατάσταση για να έχουμε αξιόπιστα στοιχεία, αλλά έχουμε στοιχεία και από άλλε πηγέ, από μη κυβερνητικέ ε, ε, οργανώσεις, όπως επίσης και από το Watch για τη Δυτική Σαχάρα. Η διαδικασία συνεχίζεται. Μπορεί να βελτιωθεί ακόμα. Η συμφωνία προβλέπει να συνεχιστούν οι ανταλλαγές μεταξύ των δύο πλευρών για να υπάρξει αξιολόγηση του αντικτύπου και να δούμε τι μέτρα θα έπρεπε να πάρουμε δεχομένω. Ξέρω ότι πολλοί από εσά ανησυχούσατε, αλλά έτσι κι αλλιώς να ξέρετε ότι δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδικασίας. Παρακολουθούμε την κατάσταση επιτόπου. Σε λίγες μέρες, αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πάει στη Δυτική Σαχάρα. Και είμαι πεπισμένος ότι θα επιβεβαιώσει τα συμπεράσματα της έκθεσης που μιλούν για σαφή ωφέλη της Δυτικής Σαχάρας. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε πριν φτάσουμε στην έγκριση της συμφωνίας. Πάντως, αναβολή για τουλάχιστον ένα χρόνο με συνέπειες νομικές που δεν θα αλλάξουν πολιτικά σημαίνει άρνηση. Αναβολή σημαίνει άρνηση ουσιαστικά. Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Θα ήταν θλιβερό. Γιατί έτσι θα παρέμενε η οικονομική αδυναμία σε βάρος της Δυτικής Σαχάρας. Τρίτο, για το σεβασμό της πολιτικής διαδικασίας του ΟΗΕ. Η συμφωνία σύνδεσης με τίποτα δεν σημαίνει ε, έμεσα αναγνώριση της Δυτικής Σαχάρας. Η πρότασή μας είναι μια τεχνική απάντηση εμπορικού χαρακτήρα και διάστασης βάσει της απόφασης του 2016 ώστε η Δυτική Σαχάρα και ο πληθυσμός της να μπορεί να υποφεληθεί από δασμολογικές προτιμήσεις. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε για το ότι θα πρέπει να συνεχίσει να υποφελείται από αυτές τις προτιμήσεις η Δυτική Σαχάρα. Όμως η Κομισιόν στηρίζει τη διαδικασία του ΟΗΕ προκειμένου να, βρεθεί, να ξεβρεθεί πολιτική λύση διαρκείας. Δύο φορές συναντήθηκα με τον κύριο Κολέρ, που είναι εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Δυτική Σαχάρα, υποσταλμένος του, και τονίσαμε ξανά και ξανά ότι στηρίζουμε τη διαδικασία του ΟΗΕ. Πρέπει να βρεθεί πολιτική λύση. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό αυτό από την εμπορική συμφωνία και σας παρακαλώ και εσάς να διατηρήσετε αυτή τη διάκριση ανάμεσα στα δύο. Γιατί αλλιώ καταλήγουμε σε ομοιρία, αν τα συνδέσουμε. Ομοιρία της μιας ή της άλλης διάστασης από την άλλη. Οπότε, υποφελούμε από την ευκαιρία που έχω σήμερα, Πρόεδρε, να σας τα διευκρινίσω όλα αυτά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λοιπόν, καλείται να αποφασίσει γνωρίζοντας συγκεκριμένα τι συμβαίνει και τι σημαίνει η τροποποίηση της συμφωνίας με το Μαρόκο. Κανείς δεν αρνείται το γεγονός ότι είναι περίπλοκη η κατάσταση, η πολιτική εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι καινούριο το ζήτημα. Σίγουρα ε, η υποστολή θα φέρει και νέα στοιχεία. Πάντως γρήγορα θα έρθει η στιγμή της πολιτικής απόφασης και το λέω και πάλι με κάθε σεβασμό, δεν σας ζητάει κανείς να αποφανθείτε για το τελικό καθεστώς της Δυτικής Σαχάρας. Κανείς. Αυτό που λέει το δικαστήριο είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια νομική βάση για να δοθεί η δασμολογική προτίμηση στα προϊόντα της Δυτικής Σαχάρας υπέρ του ντόπιου πληθυσμού. Είναι θέμα οικονομικό και κοινωνικό για την περιοχή. Θα ενισχύσει τη σταθερότητα στην περιοχή. Η συμφωνία λοιπόν, στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο στις 16 Ιουλίου, είναι μια συμφωνία στην οποία κατέληξε μετά από πολύ προσεκτική μελέτη. Τις επόμενες εβδομάδες οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ε, ε υπηρεσίας εξωτερικής δράσης θα μπορέσουν να σας προσφέρουν ό,τι οι άλλες πληροφορίες θέλετε, πραγματογνωμοσύνη και οτιδήποτε άλλο προκειμένου να αποφασίσετε. Είμαι πεπισμένος ότι τόσο θα σας πούν, θα συγκλίνουν με αυτά που σας είπα και εγώ. Ωραία, τώρα, ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, είμαι στη διάθεσή σας για αυτή την υπόθεση που είναι πολιτικά πολύ περίπλοκη, πολύ ευαίσθητη, αλλά που πρέπει να εξετάσουμε λαμβάνοντας υπόψη μας όλες τις πτυχές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μοσκόβηση. Σας ευχαριστούμε που αναφερθήκατε στα τρία αυτά ζητήματα, τα καυτά. Τώρα. Η κυρία Λαλόντ, που είναι η συγγήτρια. Παρακαλώ, κυρία Λαλόντ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, που είστε εδώ για να ανταλλάξετε απόψεις με τους ε, Ευρωπαίους Βουλευτές για αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα. Μία πρώτη ερώτηση για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα σχετικά με την επιβεβαίωση των, της ε, προέλευσης ε, των προϊόντων από την Δυτική Σαχάρα. Όπως υπόθηκε και σε προηγούμενη ανταλλαγή απόψεων, δεν υπάρχει οργανισμός ή θεσμός που, θα, που έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την προέλευση προϊόντων από τη Δυτική Σαχάρα και επομένως ε, οι μαρκινές αρχές είναι αυτές οι οποίες θα αναλάβουν το θέμα αυτό. Επομένως, το πρώτο που πρέπει να έχουμε ε, για να ε, ε, πιστοποιήσουμε ε, ότι ε, πραγματικά ε, ο πληθυσμός της Δυτικής Σαχάρας επωφελείται από τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να υπάρχει επιστοποίηση ενδεχομένως ένας τελωνιακός κώδικας για τα προϊόντα αυτά. Προτίθεστε να συνεργαστείτε με τα τελωνία κατά αυτή την έννοια ή θα δημιουργήσετε κάτι ανάλογο με τις ΗΠΑ και τις χώρες ΕΖΕΣ που έχουν αυτόν τον διαχωρισμό. Επίσης, ποιες θα ήταν οι ε, επιπτώσεις σε περίπτωση που το Κοινοβούλιο δεν επικυρώσει τη συμφωνία αυτή, δηλαδή τι μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν εάν επιβεβαιωθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ευχαριστώ σας, ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Σκιώδης ε, εισηγητές τώρα, δύο λεπτά ο καθένας. Ε, ο κύριος Σαλβατόρε Κίκου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Εγώ συμμερίζομαι τα όσα υπογράμμισε ο κύριος Επίτροπος, δηλαδή υπάρχουν δύο διαφορετικά θέματα. Υπάρχουν αυτά τα οποία αφορούν την αναγνώριση ε, θεσμική, πολιτική ε, και τα λοιπά, ε, γεωγραφική αναγνώριση και υπάρχει ένα άλλο θέμα που αφορά την εμπορική συμφωνία. Πιστεύω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι ακούστηκαν κάποιες επικριτικές φωνές όσον αφορά ακριβώς την επιβεβαίωση των ε, εκπροσώπων των φορέων, ε, των αναφορών, των οργανισμών της Δυτικής ε, Σαχάρας που δεν αναγνωρίζουν αυτούς σε σχέση με τις μαροκινές αρχές και τις, τα μαροκινά θεσμικά όργανα. Επομένως, ε, ε, θα πρέπει να ε, ενεργήσουμε με τρόπο ώστε να, να παραμείνουμε στα πλαίσια της απόφασης του δικαστηρίου. Και εδώ θα προσυπογράψω και τις ερωτήσεις της εισηγητρίας, γιατί είναι πολύ σημαντικό επί της ουσίας να κατανοήσουμε πώς θα γίνει η ταυτοποίηση της προέλευσης, πώς θα γίνει η αναγνώριση και πώς θα ε, αντιμετωπιστεί και θα προστατευτεί γενικά ε, η ε, προέλευση. Επίσης, εγώ εκπροσωπώ τη Σικελία και τη Σαρδινία και δεν πρέπει να διαπράξουμε το σφάλμα στην διαπραγμάτευση να περιλάβουμε προϊόντα τα οποία ως συνήθως θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τον νότο. Ε, γιατί μετά θα οδηγηθούμε σε μία κρίση ε, της ε, αγοράς. Θα πρέπει δηλαδή να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά αυτήν την προβληματική. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπος των σοσιαλιστών δεν είναι εδώ και επομένως θα δώσω το λόγο στον κύριο Σάντερ Λούνες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν έχω ειδική ερώτηση για τον Επίτροπο, αλλά κάτι γενικότερο να πω από πλευράς της ομάδας μου. Είχαμε το, την επιστολή σας του Αυγούστου, Πρόεδρε, και πρέπει να τη λάβουμε υπόψη. Και επίσης να ευχαριστήσουμε τον κύριο Επίτροπο που επικεντρώνεται στην νομική πτυχή, την οικονομική πτυχή και όχι τόσο στην πολιτική πτυχή της συζήτησης. Κατόπιν τούτον όμως, η ομάδα μου συμφωνεί με τον Επίτροπο ότι πρέπει να σεβόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μαρόκο. Εμείς στηρίζουμε τις προσπάθειες που κάνουν από πλευρά του ΟΗΕ. Οι ειδικοί και επεσταλμένοι, προκειμένου να βρεθεί μια βιώσιμη πολιτική λύση. Θα μελετήσουμε την νομική άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα δούμε τελικά τι θα γίνει με αυτή την συμφωνία προκειμένου να κλείσει. Ευχαριστούμε η κυρία Ρενά. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε για τις επεξηγήσεις που μας δόθηκαν. Ωστόσο, Λυπούμαστε γιατί αν βρισκόμαστε σήμερα εδώ, δηλαδή με μία απόφαση του Ευρωπαϊκού ε, Δικαστηρίου και ε, άλλες ε, αποφάσεις, είναι γιατί η εν μέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε τη δουλειά που έπρεπε να κάνει και ακριβώς επειδή υπήρχε η απόφαση του, του ε, ε, δικαστηρίου ε, καλούμαστε να τροποποιήσουμε μια συμφωνία η οποία από την αρχή θα έπρεπε να είχε λάβει υπόψη την, το καθεστώς μία αυτονομίας της Δυτικής Σαχάρας. Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να είχε δείξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεγαλύτερη δημιουργικότητα έτσι ώστε να ταυτοποιήσει τα προϊόντα της Δυτικής Σαχάρας ε, και ε, ε, επομένως να μην βάλει στο ίδιο καλάθι τα προϊόντα αυτά με τα προϊόντα του Μαρόκου. Το ξέρουμε από την αρχή το έκανε. Εν πάση περιπτώσει τώρα έχουμε μία απόφαση που λέει ότι θα πρέπει να καθοριστεί το όφελος του πληθυσμού και επίσης και κατά προτίμηση η συνένεση του, των ε, πολιτών. Ε, συμφωνώ μαζί σα ότι είναι δύσκολο, λαμβάνοντα υπόψη την ε, κατάσταση που επικρατεί, να πιστοποιήσουμε, να επιβεβαιώσουμε την συνένεση του πληθυσμού και κυρίως και γιατί γνωρίζουμε ότι το μέτωπο Πολυσάριο δεν συμφώνησε. Εν πάση περιπτώσει, το ε, γεγονός ότι δεν παρίσταται έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει κάποιο πρόβλημα είναι γεγονός ότι προκαλεί ε, πρόβλημα. Υπάρχουν όμως και άλλα προβλήματα. Προϊόντα από την Δυτική Σαχάρα πρέπει να ωφεληθούν από συγκεκριμένες ε, ελαφρύνσεις όπως και προϊόντα από το Μαρόκο αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να ταυτοποιηθούν τα προϊόντα αυτά. Εάν δεν ταυτοποιηθούν οι ε, μαροκινές αρχές ε, θα τα θεωρήσουν προϊόντα του Μαρόκου γιατί σύμφωνα με τις μαροκινές αρχές και κατανοώ τη θέση τους δεν μπορεί να πει ότι η Δυτική Σαχάρα δεν είναι μαροκινή Σαχάρα. Ε, λέμε ότι δεν θέλουμε να μπούμε στα πολιτικά ζητήματα, αλλά δεν μπορούμε να πιέσουμε το Μαρόκο να αναγνωρίσει τα προϊόντα αυτά ως μη προερχόμενα από το Μαρόκο. Εάν θέλουμε όμως εμείς να ε, σεβαστούμε το δικό μας νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή την πρόσβαση ε, σε συγκεκριμένους δασμούς, θα πρέπει να υλοποιήσουμε ε, μηχανισμούς ταυτοποίησης και διαφοροποίησης των προϊόντων αυτών. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε ότι εδώ είχαμε ήδη συμφωνίες που ε, δεν προέβλεπαν τα πάντα, ε, αλλά με καλή θέληση και του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του, ε, της Κομισιόν προσθέσαμε στις συμφωνίες αυτές κάποια πρωτόκολλα. Ζητώ λοιπόν ένα πρωτόκολλο που πριν από την κύρωση από πλευρά του Κοινοβουλίου θα καθορίζει την προέλευση των προϊόντων αυτών. Νομίζω ότι αυτή θα είναι η μόνη διέξοδος ε, που θα μας επιτρέψει σαν Κοινοβούλιο να επικυρώσουμε και τη συμφωνία ε, στην οποία έχει καταλήξει με τις Μαροκινές Αρχές. Ευχαριστώ. Κύριε Μινέρ, ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή είπε ότι η ελευτική συμφωνία με το Μαρόκο δεν μπορεί να ισχύσει στη Δυτική Σαχάρα, δεδομένου ότι δεν έχει συμφωνήσει με αυτό το τοπικός πληθυσμό. όμως τον Ιούλιο το Συμβούλιο αποφασίζει κάτι διαφορετικό. Το Πολυσάριο, που είναι ο νόμος εκπρόσωπος του λαού της Δυτικής Σαχάρας, αντέδρασε και είναι παράδοξο γιατί δεν έχει συμμετάσχει το Πολυσάριο στην απόφαση. Ενώ είναι ο νόμος εκπρόσωπος. Αν δεν συμφωνήσει το Πολυσάριο, δεν μπορούμε να αποφανθούμε ότι έχει όφελος ο πληθυσμός της Δυτικής Σαχάρας. Ελπίζω αυτή η διάσταση να συμπεριληφθεί στο κείμενο στο οποίο θα καταλήξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχω κάποιες παρατηρήσεις και εγώ μετά την παρέμβαση του Επιτρόπου του κ. Μοσκοβισή σε μια υπόθεση η οποία, όπως υπενθύμησε και ο Επίτροπος, είναι καταρχήν εμπορικός φάκελος, τεχνικός, που δεν επιδέχεται πολιτικές ερμηνείες. Το είπαμε, το έχουμε ξαναπεί κι αλλού. Υπάρχει μια διαδικασία του ΟΙΕ που συνεχίζεται για να ταυτοποιηθεί το θέμα 70 ετών πια ανάμεσα στο Πολυσάριο και το Βασίλειο του Μαρόκο και καλό θα ήταν να επικεντρωθούμε εμείς στη Δυτική Σαχάρα. Και την εμπορική αυτή συμφωνία ανάμεσα την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Σαχάρα και στα ωφέλη για τον πληθυσμό Σαχαραή που θα μπορούσε να έχει στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας και αυτού του εμπορικού πρωτοκόλου. Τα οικονομικά ωφέλη είναι σημαντικό να τα ξέρουμε. Τη απουσία δασμολογικών προτιμήσεων, οι εξαγωγές θα ήταν 6,6 εκατομμύρια σε τέλη. Κάτι το οποίο πλήττει πάρα πολύ την οικονομία της περιοχής και εμποδίζει την ανάπτυξη. Συνεπώς, το εμπόριο της Δυτικής Σαχάρας με την Ευρώπη αποτελεί και ένα μοχλό ανάπτυξης και αυτό πρέπει να το ξέρουμε θα τα δει αυτά και η αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας που θα πάει για να δει τι έχει οικοδομηθεί, τι προγράμματα γίνονται. 46,5 εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί στον πουστού για να πάρουμε το παράδειγμα της πόλης αυτής, για να υπάρξουν έργα υδροαγροτικά, ανάπτυξη της γεωργίας και εξαγωγές. Είναι πράγματα από τα οποία αναπτύσσεται η Δυτική Σαχάρα και ο λαός της. Ευχαριστούμε, Κλάος Μπούχνερ, εκ μέρους των Πρασίνων, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Με αυτή τη συμφωνία δεν εφαρμόζεται η απόφαση του δικαστηρίου γιατί έλεγε σαφώς ότι θα έπρεπε να γίνουν διαπραγματεύσεις με το λαό της Σαχάρας, ενώ εσείς κάνατε διαπραγματεύσεις με τους κατακτητές, την κυβέρνηση του Μαρόκου. Μιλήσατε με πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις, αλλά είναι χαρακτηριστικό που είπατε ότι ανα πάσα στιγμή μπορούν να μιλήσουν. Δεν είχε πει έτσι το δικαστήριο όμως την απόφασή του. Η απόφαση λέει ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνουν με κίνους, Όχι ότι ανα πάσα στιγμή μπορούν να σχολιάσουν. Κάτι άλλο σημαντικό στην απόφαση του δικαστηρίου ήταν ότι πρέπει να ωφεληθεί ο λαός των Σαχράβης εσείς. Έτσι όπως το λέτε, ο κατακτητής ωφελείται που αυτή τη στιγμή αποτελεί την πλειοψηφία του πληθυσμού. Άρα λοιπόν ε, προάγεται και βοηθάτε τους κατακτητές. Η Ισαγράβη είναι μια μειοψηφία που δεν ωφελείται και πολύ από την εμπορική συμφωνία που προωθείτε, Άρα λοιπόν η πολιτική της Ένωσης και ειδικότερα της Κομισιόν υποστηρίζει πάρα πολύ τους κατακτητές. Θυμίζω δε ότι οι ίδιοι οι Σαχράβης ε, καταπιέζονται, βασανίζονται, πρόκειται για τα χειρότερα βασανιστήρια που έχω ακούσει και ήμουν πολύ καιρό δραστηριο στη Διεθνή Αμνηστία, αυτή, αυτή ήταν η χειρότερη. Και αυτά προωθεί η Κομισιόν. Νομίζω ότι πρέπει να ντρεπόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο που ήρθε εδώ για να μιλήσει για ένα θέμα τόσο σημαντικό. Είναι δύσκολο το θέμα, θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά εδώ τα πράγματα τα κάνουμε ακόμα πιο δύσκολα. Πρώτη ερώτηση λοιπόν που σας υποβάλλω. Εκπλήσωμε, εκπλήσωμε με όλα αυτά. Γιατί έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κάνει μια συμφωνία με το Μαρόκο για την ε, Δυτική ε, Σαχάρα χωρίς όμως να έχει μιλήσει με τη Δυτική Σαχάρα, χωρίς να έχει, βάλει το πόδι, να έχει πατήσει το πόδι της στη Δυτική Σαχάρα. Ε, και ενώ αναγνωρίζει ότι δεν έχει εθνική κυριαρχία το Μαρόκο στη Δυτική Σαχάρα. Ταυτοχρόνω, η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι δεν έχει πραγματικά αριθμητικά στοιχεία σχετικά με το εμπόριο. Νομίζω ότι είναι η πρώτη και μόνη εμπορική συμφωνία που έχει υπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τέτοιε συνθήκε η Δυτική Σαχάρα, συμφωνώ μαζί σας, ότι θα πρέπει να βρεθεί το επίκεντρο όλων αυτών. Ε, όχι μόνο ε, στα, στα πλαίσια και σε σχέση με το Μαρόκο, αλλά η ίδια η Δυτική Σαχάρα. Τι κάνετε με το μη κατεχόμενο τμήμα της Δυτικής Σαχάρα, γιατί και αυτοί ε, παράγουν. η συμφωνία προβλέπεται και για αυτού, Έχετε διαπραγματευτεί με το, θέμα, με το τμήμα αυτό. Αφορά και τους δεσμεύει ή μονάχα αναφέρεστε συμφωνείτε μονάχα ε, με, την, ε, με τους κατακτητές. Επίσης λέτε ε, θα είναι μεγάλο το κόστος εάν περιμένουμε ένα χρόνο. Εγώ αντιστρέφω την ερώτηση. Ε, ποιο ε, είναι το τίμημα εάν κάνουμε κάτι που δεν είναι νόμιμο. Ε, ε, εντάξει, εσείς, εμείς λέμε ότι αυτό δεν είναι νόμιμο. Εδώ και 15, μέρες, 15 χρόνια όμως οι υπηρεσίες σας λένε ότι είναι νόμιμο. Ενώ τώρα έχουμε πλέον και την δήλωση του δικαστηρίου ότι δεν είναι νόμιμο. Ε, γιατί διαφορετικά θα φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου ε, το δικαστήριο θα ξαναπεί ότι κάτι τέτοιο δεν είναι νόμιμο και επομένως θα υποστεί σημαντικό πλήγμα η ευρωπαϊκή αξιοπιστία. Εδώ κλείνω, λέει ο Πρόεδρος, το ε, κατάλογο των αγορητών. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Στα γρήγορα μια ερώτηση. Ε, είναι δύσκολο να με πολιτική και οικονομία και, να, και τα τεχνικά νομικά θέματα. Δεν ξέρω στις διεθνείς σχέσεις ε, μπορεί αυτό να γίνεται. Είπατε, Επίτροπε, ότι δεν είναι καλό να ρωτάμε ε, το δικαστήριο αν κάτι είναι σωστό ή όχι. Ε, βέβαια, και ότι αυτό, αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει σε στάση αρνητική. Γιατί, επειδή θα το έχει απορρίψει το δικαστήριο, αλλά άμα είναι νομικό το θέμα μπορούμε να ρωτήσουμε το δικαστήριο αν οι προϋποθέσεις πληρούνται ή μπορεί να είναι ένα πολιτικό το θέμα και να μην χρειάζεται η προσφυγή εκεί. Ευχαριστώ. Γεια, Έλενα. Ναι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Επίτροπο ε, που ήρθε σήμερα ε, εδώ και Κύριε Επίτροπε, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ περίπλοκο το ζήτημα και πολύ αμφιλεγόμενο. Ε, στην ουσία, στο τέλος, ε, είναι πολιτική απόφαση, αλλά ε, είναι αλήθεια ότι θέλουν να γνωρίζουν οι βουλευτές, γυναίκες και άνδρες ε, όλα τα στοιχεία πριν πάρουν κάποια απόφαση. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερες, ε, χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες. Εγώ έχω πιστεί από αυτά που ε, λέτε, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε, και ξέρω ότι είναι πεπισμένη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να πείσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περισσότερο κόσμο. Και όπως είπε και η Μαρία Ρενά προηγουμένως, Ωστόσο, θα πρέπει να δείξει και η Κομισιόν μεγαλύτερη δημιουργικότητα έτσι ώστε ε, να ενισχύσει τη θέση της ε, με τη σύμφωνη γνώμη και άλλων. Πρόκειται για μια παγωμένη ε, σύραξη ας πούμε και εδώ όμως το Κοινοβούλιο καλείται να αποφασίσει, βρίσκεται στη μέση όλου αυτού του ζητήματος. Υπάρχουν και βουλευτές οι οποίοι θα μπορούσαν καταρχήν να συμφωνήσουν με την ανανέωση της συμφωνίας, αλλά θα πρέπει να πιστούν. Θέλουν, θέλουν όμως και όπως θέλουμε και οι περισσότεροι εδώ στο Κοινοβούλιο περισσότερα στοιχεία, περισσότερα δεδομένα γιατί βεβαίως εμείς δεν θέλουμε να αντιταχθούμε στην απόφαση του δικαστηρίου υπάρχουν, ε, ε, ε, μπορεί να περιλαμβάνει πολλά αμφιλεγόμενα στοιχεία, αλλά παρόλα αυτά είναι μια απόφαση δικαστηρίου. Γι' αυτό λοιπόν Ευχαριστούμε που είστε σήμερα εδώ. Ε, δείχνουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στην εργασία που έχετε κάνει. Αλλά μερικέ φορέ ε, για να επιτευχθεί η πλειοψηφία ε, και προκειμένου πλειοψηφία για την ανανέωση τη συμφωνία χρειάζεται μεγαλύτερη πλειοψηφία. Γιατί διαφορετικά τελικά μπορεί να φτάσουμε σε μία απόφαση και σε μία κατάσταση η οποία είναι, θα είναι κατά των συμφερόντων ε, της, ε, της Δυτικής Σαχάρας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο Μοσκοβισή που ήρθε σήμερα. Η διαδικασία διαβουλεύσεων, κεντρικό κομμάτι αυτής της ε, πρότασης, επεκρίθη πολύ όπως είπαν κι άλλοι. Εγώ θα είμαι σύντομος. Συμφωνείτε ότι η διαδικασία διαβουλεύσεων μπορεί να ισοδυναμεί με συνένεση των ανθρώπων στη Δυτική Σαχάρα αφού δεν έχει ληφθεί η άποψή τους απόλυτα. Επίσης όταν μιλάμε για ωφέλη όπως ε, είπε ο Επίτροπος από τη Συμφωνία η Επιτροπή εξέτασε τα ωφέλη και για τους Σαχράβοι που ζουν στους καταβλισμούς για τους πρόσφυγες. Επίσης πώς ε, ε, λέτε ότι είναι πολλά τα τεχνικά θέματα αλλά η διαδικασία που ακολουθήθηκε εδώ και δεκαετίες δεν έδωσε αποτελέσματα. Είναι σταγόνα στον ωκεανό ή στην έρημο. Πρέπει λοιπόν να μας πείτε ε, τι, πώς αντιμετωπίζεται η πολιτική πραγματικότητα με το έργο του, των Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Μοσκοβισή για το όσο μας είπε. Μια σύντομη ερώτηση, μια διευκρίνηση. Συμφωνώ ότι οι όροι έχουν πολύ μεγάλη σημασία για να καταλαβαίνόμαστε όταν μιλάμε. Κυρίως όταν πρόκειται για νομικά ζητήματα που διακρίνονται από τα πολιτικά. Γι' αυτό και με εκπλήσει που μιλάτε για διαβούλευση. Μα η απόφαση του δικαστηρίου δεν μιλάει για διαβούλευση, μιλάει για συνένεση καταλαβαίνετε ότι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ούτε μιλάει για τον τοπικό πληθυσμό. Μιλάει για τον πληθυσμό Σαχαραουή και ο ΙΕ. Και εδώ δεν μιλάω για κανέναν ύποπτο, καμιά ύποπτη οργάνωση που τη θεωρεί έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλάει για τον Λό Σαχαροή, αναγνωρίζεται ότι, ο νο... ότι η η δομή η οποία νόμιμα εκπροσωπεί τον λαό Σαχαροή είναι το μέτωπο Πολυσάριο. Τελείωσε. Αυτά ήθελα να διευκρινίσω, γιατί είναι σημαντικό η ορολογία και το θέμα το άλλο. Τώρα εντάξει, δεν θα πρέπει ίσω να μπούμε σε πολιτικά ζητήματα, αλλά μια που είμαι κοινοβουλευτική εκπρόσωπο, θέλω να σα πω το εξή. Αναρωτιέμαι, γιατί γίνεται συμφωνία με το Μαρόκο που είναι κατοχική δύναμη και δεν γίνεται με την διοικητική δύναμη που είναι η Ισπανία, κάντε τη συμφωνία με την Ισπανία και όχι με το Μαρόκο. Η κυρία Χαουτάλα. Ευχαριστώ πολύ. Επίτροπε, οι υπηρεσίες σας εξέδωσαν σημείωμα φέτος το Φεβρουάριο στα κράτη-μέλη, στις θελωνιακές τους αρχές και τους είπατε ότι πρέπει να γίνονται κατασχέσεις μαροκινών εμπορευμάτων αν υπάρχει αμφιβολία για την ε, καταγωγή των εμπορευμάτων από την Δυτική Σαχάρα. Και οι συνάδελφοι συνάντησαν το Μαροκινό Γραφείο Εμπορίου και τους είπαν ότι συστηματικά αρνούνται να αναφέρουν τη Δυτική Σαχάρα ως ε, περιοχή καταγωγής των προϊόντων. Οι οδηγίες σας λοιπόν θα ε, λύσουν το πρόβλημα στη συνεργασία ε, των τελωνιακών αρχών. Υπάρχουν πολλά θέματα εδώ νομικά. Μπορείτε να κάνετε μια σύγκριση, ας πούμε, γιατί η κατάσταση μεταξύ Μαρόκου και Δυτικής Σαχάρας είναι διαφορετική σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, αντίθετη από τις σχέσεις Ρωσίας-Κρυμαίας. Και τέλος, η πρόεδρος της αντιπροσωπείας με το Μαγκρέμπ, η κυρία Ινέσα Γιάλα Ζέντερ. Ευχαριστώ πολύ. Άργησα γιατί είχα άλλα θέματα και δεν άκουσα όσα είπε ο Επίτροπος, αλλά στην αντιπροσωπή για το Μαγκρέπ παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά όλες τις προσπάθειες που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση ακριβώς με την αναγκαιότητα αυτή να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που θέτει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Είναι αλήθεια ότι όπως είπε και η κυρία Βαλενθιάνο έχει κάποιες ε, πτυχές που θα έπρεπε να τους ρωτήσουμε. Δηλαδή πώς θεωρεί το δικαστήριο ότι επιτυχάνεται η συνένεση του πληθυσμού. Κάτι με το οποίο έτσι κι αλλιώ ε, θα έπρεπε να είχαμε ξεμπερδέψει τόσα χρόνια που δουλεύει πάνω σε αυτό ο ΙΕ. Πάντω το θέμα των ε, βοηθειών και του προπολογισμού δεν έχει λυθεί ακριβώς γιατί ο ΙΕ δεν έχει καταλήξει, δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι σήμερα βρισκόμαστε ως Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο στη μέση και εμείς πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε να συνδυάσουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Τα ξέρουμε και ακούγονται. Δεν πρόκειται για απειλή, αλλά πρόκειται για μια πραγματικότητα συγκεκριμένη που έχουμε επιτόπου. Και συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να βρει τον τρίτο δρόμο, την ανατολική διαδρομή, έτσι ώστε να μπορέσουν να φτάσουν εκείνοι που δεν μπορούν να μπουν από τους άλλους δύο δρόμους. Κάτι το οποίο καταστρέφει μια περίπλοκη οικονομία που έχει βέβαια τα προβλήματά της, η Μαροκινή. Να αναγνωρίσουμε όμως τα δικαιώματα, κάτι το οποίο Προσπάθησε να πετύχει η Επιτροπή με την διαβούλευση, αλλά να ξέρουμε ότι η Σαραουή δεν είναι μόνο κάτι ενιαίο, υπάρχουν πολλοί και διάφοροι. Τα ξέρουμε. Ήρθε και πρόεδρος του Πολυσάριου που τον έχουν εκλέξει δική του. Είχαμε σχέσεις με όλους αυτούς, με τους οποίους μίλησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους ρώτησε, τους τη γνώμη τους. Οπότε συμφωνούμε ότι πρέπει να στηριχτεί η πρόταση. Αναγνωρίζω ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, αλλά το πρόβλημα είναι να δούμε πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καταφέρει να συμφωνήσει για το τι ισχύει σε μια περιοχή όπου μπλέκονται δύο χώρες, γιατί υπάρχει και Αλγερία, μην το ξεχνάμε, έτσι. Είναι κάτι που πρέπει να λύσουμε εμείς. Εδώ δεν το έχει λύσει ο ΙΕ τόσα χρόνια. Θα πρέπει πάντως να εμπιστευτούμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λύσει ένα πρόβλημα που δεν δημιουργήσαμε εμείς. Κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ. Η συζήτηση η οποία έλαβε χώρα ακριβώς καταδεικνύει την πολιτική, νομική και γενική περιπλοκότητα ε, του ε, θέματος ε, αυτού. Είναι δύσκολο όντω να μην υπάρχει καμία πολιτική χρειά στο όλο θέμα του του λεχθέντος πάντως. Η Κομισιόν προσπάθησε έτσι ώστε η απάντηση να είναι όσο γίνεται περισσότερο νομική ε, και οικονομική σε ένα νομικό πρόβλημα. Ε, ίσως σας απογοητεύσω, αλλά δεν θέλω να ε, μπω στην γεωπολιτική ή στρατηγική συζήτηση, άλλωστε δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητος. Αυτό ακριβώς θέλαμε να αποφύγουμε άλλωστε στην προσέγγιση την οποία επιλέξαμε στα πλαίσια της συμμόρφωσης με μία νομική απόφαση και το θέμα του καταστατικού ε, ε, και του καθεστώτος ε, της Δυτικής Σαχάρας δεν μπορεί να μας απασχολήσει ακριβώς εδώ. Ναι, Βεβαίως ε, εγώ αντιπαρέρχομαι ε, κάποιες ε, απολύτως λανθασμένες τοποθετήσεις οι οποίες εν παρόδο ανεφέρθησαν ότι δήθεν η Κομισιόν παραβλέπει ή και υποστηρίζει κάποιες, κάποια βασανιστήρια και τέτοιου είδους πρακτικές. Αυτό βεβαίως δεν ισχύει. Εγώ κατανοώ ότι χρειάζεστε ίσως ε, κάποια στοιχεία εμβάθυνσης ε, πριν πάρετε την απόφασή σας. Ε, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω και σας το υπογράφω είναι ότι η συζήτηση και η εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπήρξε εργόδης και υπήρξε μακρόχρονη. Και βεβαίως εγώ είμαι απολύτως διατεθειμένος να επανέλθω ε, μετά την αποστολή ε, επιτόπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να ανταλλάξουμε περαιτέρω απόψεις. Νομίζω ότι μπορούμε να ε, προοδεύσουμε στη συζήτηση, να προχωρήσουμε στη συζήτηση με τον τρόπο αυτό. Αλλά πιστεύω ότι η πρόταση έχει υποστεί τόσο σοβαρή επεξεργασία ώστε να είστε σε θέση να την δεχτείτε. Τρίτη παρατήρηση εισαγωγική κατά κάποιο τρόπο. Ας αποφύγουμε να θέσουμε σαν ε, προηγούμενο και σαν προαπαιτούμενο την επίλυση της ε, κατάστασης έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην συζήτηση αυτή. Αλλά βεβαίως μπορώ να κάνω και κάποιες εκτιμήσεις για συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν και από την εισηγήτρια και από σκιώδεις εισηγητές. Πρώτον, όσον αφορά ε, τα θέματα ε, της επιβεβαιωμένης προέλευσης από τη Δυτική Σαχάρα. Για να μπορέσουμε να έχουμε τη βεβαιότητα ότι επωφελείται ο τοπικός ε, πληθυσμός και η κοινότητα ε, από την ε, συμφωνία ναι, θα χρειαστεί η, μέγιστη, η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια. Αλλά Βεβαίω, καταλαβαίνετε ότι ξεκινάει ένα φαύρο κύκλο όσον αφορά τη δυνατότητα ταυτοποίηση επίσημη των προϊόντων αυτών. Ωστόσο, υπάρχει μια ομάδα η οποία εργάζεται πάνω, στο θέμα, πάνω στα θέματα αυτά να σας πω ότι υπάρχουν και προς του Μαρόκου που συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή και εν πάση περιπτώσει πρόκειται για ένα θέμα επί του οποίου ε, ε, ε, είμαστε ήδη αλλά θα είμαστε και στο μέλλον εξαιρετικά απαιτητικοί οπωσδήποτε θα ανταλλάσσονται πληροφορίες ε, ε, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ε, σύμφωνα με τις διαδικασίες της Συμφωνίας Σύνδεσης. Επίσης σε υπουργικό επίπεδο έχουμε συγκεκριμένες επαφές με το Μαρόκο και σας διαβεβαιώ ότι θα είμαστε ιδιαίτερος απαιτητικοί. Δεύτερο θέμα το οποίο έθιξαν πολύ μεταξύ ημών οι επιπτώσεις σε περίπτωση μη ε, ε, επικύρωσης της ε, συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε υποχρεωμένοι να διαπιστώσουμε ότι θα είναι σαφής οι επιπτώσεις. Δεν θα υπάρξει προτιμησιακό καθεστώς και αυτό βεβαίως θα έχει αρνητικό αντίκτυπο ε, όσον αφορά το οικονομικό όφελος της ε, ε, περιοχής και υπενθυμίζω ότι η περιοχή αυτή εξαρτάται από τη γεωργία και από την αλία. Ε, την μεταποίηση επίσης των ε, προϊόντων της ε, αλίας που ενδεχομένως η μεταποίηση αυτή ίσως είναι παράδοξο αλλά πάντως είναι πολύ πιθανό να μετακινηθεί προς το Μαρόκο πράγμα που σημαίνει ότι με κανένα τρόπο δεν θα υποστηριχθούν οι δραστηριότητες της Δυτικής Σαχάρας. Αναγνωρίζω λοιπόν ότι η Κομισιόν έκανε ό,τι μπορούσε καλύτερο και περισσότερο έτσι ώστε ε, να επιτύχει πληροφορίες, πληροφορίες οι οποίες ε, ε, εν επετέφθησαν και μέσω των σχέσεων με το Μαρόκο αλλά και από εκθέσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων κλπ. Επίσης δεν είναι δυνατόν να βασίσουμε αποφάσεις πάνω σε περιστασιακές και αποσπασματικές αναφορές. Χρειαζόμαστε διαρκή και σοβαρή πληροφόρηση. Επίσης εδώ είναι ένας φαύλος κύκλος. Είναι ποιος γέννη, αν, αν η κότα γέννησε το αυγό ή το αυγό την κότα. Αυτό που καλούμαστε εμείς να διασφαλίσουμε είναι ότι θα υπάρξουν τα, τα μέτρα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή εφαρμογή ε, του προτιμησιακού καθεστώτος, ε, δηλαδή καλή συνεργασία μεταξύ των τελωνιακών αρχών, έλεγχος, επιθεωρήσεις κλπ είναι ο μόνος τρόπος έτσι ώστε μια τέτοια συμφωνία να μπορέσει να λειτουργήσει. Ε, ε, αυτό που μας ενδιαφέρει φυσικά είναι να έχει αποτέλεσμα συγκεκριμένο, συγκεκριμένα παραδοτέα να προκύψουν από αυτήν την ε, συμφωνία και όφελος και για τη Δυτική Σαχάρα. Τώρα σε σχέση με αυτό που είπατε για την ε, ε, Σικελία και τη Σαρδινία μου φαινόταν απολύτως ε, λογικό ότι δεν θα υπάρξουν έμεσες αρνητικές επιπτώσεις για τις περιοχές αυτές. Επίσης, κατανοώ αυτό που λέει η κυρία Γιάλα Σέντερ σχετικά με την διαβούλευση και την συνένεση αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο με πολύ δύσκολο είναι ε, να ε, λυθεί. Και αυτό που προσπάθησε να κάνει η Κομισιόν είναι ε, να ε, ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ε, στο περίπλοκο αυτό πρόβλημα. Θελήσαμε να καλέσουμε τις κυριότερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κοινωνικές οργανώσεις κλπ. 25 ομάδες ή πολιτικές, πολιτικοί οικονομικοί πρωταγωνιστές που σχεδόν όλοι δέχτηκαν, αποδέχτηκαν ε, την πρόσκλησή μας. Πέντε ε, δεν ενέδωσαν στις επανειλημμένες προσκλήσεις μας. Απ' την άλλη πλευρά ε, δεν υπάρχουν ε, συγκεκριμένες αντίθετες απόψεις παρά μόνο μιας πλατφόρμας ε, όπου συγκεντρώνει διάφορες μικρές μη κυβερνητικές οργανώσεις όσον αφορά αντίθεση όσον αφορά το περιεχόμενο της ε, συμφωνίας. και νομίζω ότι αυτό καταδεικνύει ότι τουλάχιστον οι τεχνικές ε, πλευρές της συμφωνίας έχουν ε, ε, καλυφθεί. Τώρα βεβαίως το μπαλάκι είναι στην πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο θα πρέπει να ασκήσει τις δικές του δικαιοδοσίες και να δει αν μπορεί να επικυρώσει αυτήν την πρόταση. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που ήθελα να κάνω. Βεβαίω δεν παραβλέπω και δεν παραγνωρίζω καθόλου ε, τις ιδιαίτερες δυσκολίες του θέματος, τον ειδικό χαρακτήρα κτλ αλλά εγώ δεν θέλω να εμπλακώ στην επί της συζήτηση και την πολιτική συζήτηση. Έχουμε εδώ την απόφαση του δικαστηρίου. Ναι, ε, ίσως κυρία Ρενά είπατε ότι πρέπει να αποφύγουμε τέτοιου είδους ε, προσφυγές και αποφάσεις, ε, ε, αλλά η απόφαση είναι αυτή και είναι εδώ. Και άλλωστε τίποτα δεν είναι τέλειο. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, εγώ απαντώ τεχνικά και νομικά, έχοντας υπόψη μου αυτήν την απόφαση και αν θέλουμε να διασφαλιστούν ε, ε, οι οικονομικές ε, ροές και αν θέλουμε να ωφεληθεί ο πληθυσμός της Δυτικής Σαχάρας τότε θα πρέπει να ληφθούν όλα αυτά τα στοιχεία υπόψη. Και εν τέλει πιστεύω ότι η πρόταση που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια καλά προετοιμασμένη και σωστή πρόταση, είναι μια γεράχτισμένη πρόταση. και ε, ε, ξέρετε ότι οτιδήποτε δεν προχωράει στην, στις επιτόπου διαδικασίες εν τέλει στρέφεται εναντίον ή ζημιώνει τους τοπικούς ε, πληθυσμούς. Και αυτό το λαμβάνουμε εμείς υπόψη στην Κομισιόν. Όπως άλλωστε λάβαμε υπόψη όλα τα πιθανά στοιχεία τα οποία αφορούν και τη δικαιοσύνη και την οικονομία κλπ. Ε, και λέω ότι ε, εάν ξεκινήσουν ε, πάλι διαδικασίες θα έχουμε χάσει έναν ακόμα χρόνο. και ούτε όλες οι απαντήσεις ε, μπορούν να δοθούν σε μια συζήτηση την οποία σέβομαι ε, βαθύτατα. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι είμαι στη διάθεσή σας ε, έτσι ώστε να έχουμε κι άλλη ανταλλαγή απόψεων μετά από την δική σας επίσκεψη. Αλλά να σας πω ότι εμείς δουλεύουμε γιατί θέλουμε να ωφεληθούν και οι πληθυσμοί της Δυτικής Σαχάρας. Ε, με ηρεμία λοιπόν και ε, ε, γαλήνη πνεύματος σας ζητώ να υποστηρίξετε την πρόταση της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε, λέει ο Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο στην ε, εισηγήτρια, στην κυρία Λαλόν, για μια πάρα πολύ σύντομη ε, τελική ε, παρατήρηση. Ναι, πολύ σύντομη. Θα ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Επίτροπο για τις απαντήσεις που έδωσε για ένα θέμα που γνωρίζω και αναγνωρίζω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Ε, εμείς θα έχουμε σε μια εβδομάδα την αποστολή μας επί τόπου. Ελπίζω ότι θα δώσει καρπούς αυτή η αποστολή, αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και το λέω εξ αρχής να αποσυνδέσουμε εντελώς τα γεωπολιτικά από τα ε, οικονομικά και εμπορικά. Θα συζητήσουμε μετά την επίσκεψη στο Μαρόκο. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Τώρα θα αλλάξουμε αίθουσα και θα πάμε στην 2Q2, στο κτίριο Αντάλ.